Okay, good afternoon everybody. I think we can make a... Ας αρχίσουμε λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Ελπίζω ότι ξεκουραστήκατε όσοι κάνατε διακοπές, όσοι πήγατε σε αποστολές, ελπίζω οι αποστολές σας να πήγανε καλά. Ξέρω ότι είναι μια αποστολή στο Καμερούν για ζητήματα δασοκομείας και κάποιοι συναδελφοί μας είχαν πάει. Είναι πλήρη η ημερήσια διαταξή μα σήμερα και γι' αυτό θέλω να αρχίσω έγκαιρα. Πρώτο θέμα λοιπόν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε να προτείνετε αλλαγές, μπορεί να εγκριθεί ως έχει. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν. Για τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρώτη ανακοίνωση, σημαντική και για το προσωπικό. Έχουμε ψηφοφορία σήμερα στις 5 και 4. 5 και 4 για το European Consensus on Development. φροντίστε να έχετε τις κάρτες σας, γιατί καμιά φορά ορισμένοι τις ξεχνούν λοιπόν να φροντίσετε και εσείς οι ε, συνεργάτες να θυμίσετε στα μέλη να έλθουν με τις κάρτες τους στις 5 και 4. Και θα είναι ακριβώς 5 και 4 ακόμα και αν ε, τελειώσουμε νωρίτερα. Θα περιμένουμε τότε. Δηλαδή. Δεύτερη ανακοίνωση. European Development Days. Οι περισσότεροι που είστε εδώ γνωρίζετε ότι αυτές οι Development Days είναι πολύ ενδιαφέρουσες γιατί συνέρχονται μη κρατικέ οργανώσει, ε, εμπειρογνώμονε, ε, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, οι κομισιόν. Γίνονται την επόμενη εβδομάδα, 5-8 Ιουνίου, και η Επιτροπή μα την επόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη επόμενη εβδομάδα δηλαδή, και η δική μα Επιτροπή και η Επιτροπή Περιβάλλοντος διεξάγουμε ειδική συνεδρίαση για τους στόχους 2030 για την ευημερία και τους άλλους στόχους του 2030 με την ιδέα να μιλήσουμε με ειδικού εκπροσώπους του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για παράδειγμα και με τον Μποχόμοντ Γιούνους, ε, νομομαθή, δικηγόρο δηλαδή, όπως και οι άλλοι, που βρέχεται από τον Μπαγκλαντές, πολύ γνωστό πρόσωπο έχει δημιουργηθεί και με βραβείο Νόβελ, για, τις, ε, για τα ζητήματα της ανάπτυξης. Πολύ σημαντική λοιπόν η συνάντηση αυτή, θα έχουμε εξάλλου και τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας και συμπρόεδρο ίσως είναι και φιλικού γένους, ένα Σόλμπεργκ. Για την ομάδα αυτή που ασχολείται με τους ε, στόχους του 2030. Πολύ σημαντικό, 3 και 4 την επόμενη Τετάρτη 7 Ιουνίου από τις 3 και 4 μέχρι τις 4 και 30. Μία ώρα και 15 λεπτά. Έκτακτη συνεδρίαση επιτροπή Επιτροπής μας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στην διάρκεια των Development Days ε, θα έχουμε ένα πάνελ υψηλού επίπεδου που οργανώνει η Επιτροπή μας. Αυτοί οι Development Days διεξάγονται εκτός σε ένα μεγάλο κέντρο συνεδριάσεων και συνεδρίων που λέγεται Tour Taxi στις Βρυξέλλες και είναι στις 8 Ιουνίου το πρωί. Εκείνη την ημέρα βέβαια διεξάγονται οι Βρετανικές εκλογές, οπότε εγώ δεν θα είμαι παρούσα. Όμως θα είναι εδώ η Ελισλάιν, ο Μπόγκταν Βέντε και θα ηγηθούν τη συνάντηση αυτής που ασχολείται με ζητήματα μετανάστευσης. Ελπίζω ότι εσείς θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στις Development Days θα σας δώσω αμέσως το λόγο σε εσά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν γνωρίζετε πώς θα πάρετε την άδεια εσόδου, να ρωτήσετε τη γραμματεία, το badge δηλαδή. Αν θέλετε να συμμετάσχετε. Πιστεύω θα έχετε και πρόγραμμα, έτσι δεν είναι, ή των εργασιών των Development Days, γιατί θα διεξάγονται διάφορες εκδηλώσεις. Θα σας ενημερώσουμε πάντως και γραπτός. Αλλά θα δώσω αμέσως σε λίγο το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχετε ερωτήσεις? Για το 3 λοιπόν, έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων, δηλαδή της 20 και 21 Μαρτίου 2017, ως συνήθως, ό,τι παρατηρήσεις έχετε, να τις κοινοποιήσετε στη γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδριάσεως. Και αλλιώς θα θεωρηθεί, θα θεωρηθεί εγκεκριμένο το πρακτικό. Τέταρτο, ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από ό,τι μαθαίνω, ο Κάρστιν Σόρενσεν Κάστιν Σόρενσεν, έχετε κάποιε παρατηρήσει να κάνετε. Ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχα κάποιες παρατηρήσεις να υπενθυμίσω σε όλους ε, της European Development Days και ότι προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας σε αυτό το υψηλό επίπεδο ε, γεγονός ε, που θα έχει ε, πάρα πολλούς συμμετέχοντες. Ναι, όπως είπαμε, καλωσορίζουμε το Development Dates. Είναι μεγάλο ζήτημα και θα ασχοληθούμε με μεγάλα ζητήματα στον τομέα της ανάπτυξης. Ωραία, πάμε στο σημείο 5. Αντιμετώπιση της ρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Η συγγητρία είναι η Τερέσα Χιμένες Μπεθερίλ. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Ξέρουμε ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες ε, χώρες ε, υφίστανται πιέσεις οι κοινωνίε των πολιτών από τις κυβερνήσεις. Ε, ζητούν οι κυβερνήσεις από τους διεθνείς οργανισμούς να φύγουν και ασκούν πίεση στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια συνδεδεμένη επιτροπή δύναμη του άρθρου 54 γιατί έχει αρμοδιότητα και αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μεγάλο το θέμα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην εισηγητρία στην Τερέσα. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Ευχαριστώ πολύ. Στα τέλη Απριλίου είχα την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το ανησυχητικό θέμα ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, αφορούσε την παρουσίαση και τη μελέτη της Επιτροπής για το θέμα αυτό ε, δύναμη του άρθρου 54. Ένας άλλος συζητητής, ο Φραντζέσκο ε, Δρεσής, ασχολήθηκε με αυτό και συνεργαζόμαστε άριστα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Υπάρχουν κάποια θέματα που παρατηρήσαμε ότι η κοινωνία των πολιτών είναι σημαντική για την ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενε χώρε. Σε δεύτερο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζεται η καταστολή της κοινωνίας των πολιτών ε, και των οργανισμών που την εκπροσωπούν διάφοροι οργανισμοί, διαφορε πλατφόρμες πολιτών, ιδρύματα. Ήδη αυτό αιτιολογεί την ύπαρξη αυτής της ε, γνωμοδότησης, διότι υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και μας βοηθά να δούμε ποιοι οργανισμοί τις υποστηρίζουν και επίσης έχουμε και ένα αντίθετο σενάριο που αναφέρεται σε αυτή τη γνωμοδότηση, το σενάριο όπου τέτοιες οργανώσεις πέφτουν θύματα κάποιων ε, κυβερνήσεων. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά κάποιες χώρες τις θεωρούν εχθρούς τις οργανώσεις αυτές ε, ε, που προσπαθούν να καταγγέλουν ε, καταχρήσεις προς τους πολίτες και μερικές φορές είναι ο μόνος υπερασπιστής τέτοιων, ανθρώπων, τέτοιων πολιτών. Παρουσιάζω λοιπόν την έκθεση που υπάρχει ήδη σε όλες τις γλώσσες και όπου παρουσιάζω τις ανησυχίες μου και τα οραματά μου. Εγώ προέρχομαι από την κοινωνία των πολιτών η πολιτική μου συμμετοχή γεννήθηκε σε τέτοιες οργανώσεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνία των πολιτών. Ανέκαθεν ναι, υποστήριζα τα θύματα, ε, πιο συγκεκριμένα της τρομοκρατίας, ε, αλλά και άλλων ειδών θύματα. Είμαι, έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω ορισμένες παραγράφους στην ιδεολογική σκέψη G αναφέρεται η σημερινή κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών, ο μετασχηματισμός της και οι απειλές που υφίσταται. Αναγνωρίζει την καταστολή από πλευράς ορισμένων κυβερνήσεων ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Και στις δύο πρώτες παραγράφους εκφράζω αυτό που είπα αρχικά. Υπογραμμίζω δηλαδή ότι μια κοινωνία των πολιτών είναι κάτι απαραίτητο να υπάρχει ως ανεξάρτητη δομή, πλουραλιστική δομή, ε, κάτι σημαντικό για την ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας. Στη δεύτερη παράγραφο υπογραμμίζω το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες και πόσο σημαντικός είναι. Στην πέντε υπογραμμίζω τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν υπάρχουν προβλήματα όπω αυτά που αναφέρουμε για την κοινωνία των πολιτών, πρέπει να γίνουν κάποιε προσπάθειε και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό ε, ε, παράγων υπεράσπιση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη κοινωνία των πολιτών. Μέσω λοιπόν ενεργών πολιτικών, ενίσχυση τη κοινωνία των πολιτών στι αναπτυσσόμενε χώρε θα επιτευχθούν όλα αυτά. Και επιθυμίζω ότι υπάρχουν διάφορα εργαλεία όπω το Εργαλείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό Καταπίστευμα για τη Δημοκρατία που θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την κοινωνία των πολιτών σε 105 χώρες. Παρουσιάζω λοιπόν τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητώ τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη. Και όπως λέω και στις τελικές παραγράφους χρειάζεται και χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο να προωθηθεί και η συμμετοχή εξωτερικά και εσωτερικά ε, επιδιώκοντα κάποια συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη και εκτό. Εμεί είμαστε σημαντικό παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτικά είμαστε ο μεγαλύτερο χρηματοδότη, αλλά δεν λέω ότι πρέπει να παρεύουμε πολιτικά στα όσα κάνουν άλλε χώρε, αλλά δεδομένου οικονομ... της οικονομικής μας και τη οικονομική μα συμμετοχή. Στι αντιπροσωπείε μα, ε, στι άλλε χώρε αυτέ Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι γίνεται με το θέμα των προσφύγων, τι γίνεται στα σύνορα τη Συρίας. Είδα ότι στο Λίβανο, για παράδειγμα, όταν μιλάνε για του διάφορου συμμετέχοντε που κάθονται σε ένα τραπέζι για να επιλύσουν ε, το πρόβλημα του πολέμου, εκεί μιλάνε για 5-6 συμμετέχοντες, δεν αναφέρουν ποτέ την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα από του μεγαλύτερου ε, δωρητέ βοήθεια. σε επίπεδο αντιπροσωπιών, για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Πήγα στο Μεξικό και επέμεινα για να μπορέσουμε να συνεντήσουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να κάνει αντιπροσωπεία μου για το Μεξικό, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες αντιπροσωπείες. Η δική μου θέση βασίζεται στην υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών ε, για να υπάρξει μια ίση αντιμετώπιση. Σας υπενθυμίζω ότι στις 31 Μαΐου, την Τετάρτη, είναι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών και υποφελούμε της ευκαιρίας αυτής για να σας πω ότι είμαι διαθέσιμη στα μέλη της αντιπροσωπείας που θα ήθελα να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Ευχαριστώ. Ανής που αντικαθιστά τον, τον Τουρού. Ναι, πράγματι. Αντικαθιστώ την συνάδελφό μας Φουντζούλιτσα που ε, κολλείεται. Γι' αυτό να με επιτρέψει να διαβάσω ένα ε, κείμενο που μου έχει δώσει. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια όπως είπα ε, εξ ονόματος ε, της αδρού μας, που δυστυχώς κολλείται. Το σχέδιο εκθέσεως καλύπτει πολλά σημαντικά θέματα. Ο συναδελφός πιστεύει ότι ορισμένα πρέπει να ενισχυθούν από αυτά που λέει. Με τη γενική σκέψη ότι δυστυχώς όχι μόνο οι αναπτυσσόμενες χώρες περιορίζουν τον χώρο των πολιτών, αλλά και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με είναι ένα ζήτημα παγκοσμιοποίησης για να έχει αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αντιληφθεί και αυτή ότι εδώ αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και να τονίσουμε ότι χρειάζεται διάλογος μεταξύ αντιπροσδέσεων και κυβερνήσεων. Και στις εμπορικές συμφωνίες και στις εμπορικές συνεργασίες πρέπει να ενισχυθούν υπέρ της ευημερίας της κοινωνίας των πολιτών. Είναι θεμελιώδες να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των CSO που εργάζονται επί τόπου και η μείωση του πεδίου πρωτοβουλειών τους. Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί και η συνεργασία νότου-νότου, γιατί ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μπορέσει να αναπτύξουν τον χώρο όπου λειτουργούν και οι CSO, η Civil Society Organizations. Θα συνεργαστούμε βεβαίως για τη σύνταξη αυτής της σημαντικής εκθέσεως. Αυτό είναι το κείμενο του συναδέλφου μας και ήθελα επίσης και εγώ με τη σειρά μου να τονίσω ότι είναι ε, αναγκαίο, εάν εξετάσουμε δηλαδή την ορθή, τη χρηστή διακυβέρνηση, είναι σημαντικό ε, να τους ενισχύσουμε και ιδίω τους ε, στόχους που είναι σημαντικές για πολλές χώρες και στο πλαίσιο του περιορισμού του χώρου ε, δράσεως της, ε, των ε, οργανώσεων και των πολιτών. Μιλήσατε για το παρελθόν σας και εγώ μεγάλωσα σε ένα καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού. Για την Ουγγαρία λοιπόν είναι σημαντικό όπως ο περιορισμός της ελευθεροτυπίας και της πολιτιστικής ελευθερίας όπως στην Πολωνία. όπου διώχνουν ανθρώπους που διευθύνουν θέατρα και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια κλπ. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτό, πρέπει να συνδεθεί με τους ε, στόχους και να δοθεί και μια ευρωπαϊκή προοπτική. Ευχαριστώ. Γκέρενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ ε, συμφωνώ. Αντικαθιστώ εδώ τον κύριο Λουί Μισελ είναι βεβαίως δύσκολο να αντικαταστήσει κανείς τον Λουί Μισελ. Ε, μιλάω το για το χρόνο που θα του είχε δοθεί. Προτού το κάνω αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να της προτείνω ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον τίτλο της εισήγησης καταπολέμηση της συρρήκνωσης του χώρου για την κοινωνία των πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες μας επίσης θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, διότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν το παν για να δώσουν ένα συγκεκριμένο νόημα στη συρρήκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά σαφείς έτσι με αυτόν τον νέο τίτλο το κείμενο του Λουί Μισελ είναι ότι ευχαριστεί του συγγραφεί του κειμένου αυτού και νομίζω ότι, νομίζει ότι είναι καλή βάση εργασία, η κοινωνία των πολιτών και οι μη κρατικοί πρωταγωνιστές είναι σημαντικοί. Δεν χρειάζεται ο ρόλος του εταίρου για την υποβολή προγραμμάτων, αλλά η παρουσία του σε μια κοινωνία είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη, διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κοινωνία των πολιτών είναι κάτι απαραίτητο, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το ρόλο ε, του καθενός. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη τη στο λαό, η κοινωνία των πολιτών έχει συμπληρωματικά ρόλο, θα πρέπει να προωθήσει την αλλαγή της ε, προτάσεις ε, και θα είναι μια δύναμη που οδηγεί τον πολίτη να λάβει μέρος ε, στις ε, συζητήσεις για την κοινωνία, για τα κοινωνικά και τα οικονομικά θέματα. Η δυτική κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να ενισχύσει τις ΜΚΟ με τεχνογνωσία για να τις βοηθήσει με υπεύθυνο τρόπο να συμβάλλουν ε, στην ανάπτυξη της χώρας τους. Είναι μια πρόκληση σημαντική και ομολογώ, λέει ο Λουί Μισελ, ότι έχω την εντύπωση ότι αυτού του είδους της μεταφοράς δεν γίνεται με παρκή τρόπο και ότι οι δυτικές οργανώσεις ε, αντικαθιστούν πολύ συχνά την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια για την ασφάλεια, την ανάπτυξη. Οι ΜΚΟ πρέπει όχι μόνο να αναπτύσσουν αναπτυξιακά προγράμματα και να ανταποκρίνονται σε άμεσε ανάγκε. Υπενθυμίζω τον σημαντικό ρόλο τη διασπορά που έχει τα μέσα ως διεπαφή να προσφέρει πολλά στην χώρα προέλευσης. Ο Λουί Μισελ εισήγαγε τροπολογίε προ την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι η παρέμβαση του Λουί Μισελ. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Στην ε, σύμβαση του Κοτονού στι 23 Ιανουαρίου 2000 Ιουνίου ε, είχαμε προβλέψει μια διάταξη για την προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες ΑΚΕ. Η Κομισιό διαθέτει ένα, έναν απολογισμό, μια εκτίμηση, μια αξιολόγηση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της διάταξης. Ξέρω ότι τότε και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το μικρό μας δάχτυλο. Τα πάντα έγιναν από ευρωπαϊκής πλευράς για να πιστούν οι χώρες ΣΑΚΕ να δεχθούν την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες τους. Χρειάστηκε να το επιβάλλουμε αυτό. Τόσο υπήρχαν επιφυλάξεις από πλευράς των αναπτυσσομένων χωρών, αλλά νομίζω ότι μπορώ να πω με τον Λουί Μισελ και τον Ισίτη Λουίτ ότι κάτι αυτό είναι σημαντικό να έχουμε γέφυρες, να έχουμε εταίρους, να έχουμε ανταλλαγέ και να έχουμε μια σκητάλη αν θέλετε ε, αυτούς ε, που ζυμώνουν νέες ιδέες. Αυτή είναι η πρόταση. Υπάρχει καμία μελέτη αντικτύπου σχετικά με αυτή τη διάταξη που είχε εισηχθεί στη συμφωνία αυτή με τις ε, χώρες εταίρους. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θα πάρει σε λίγο το λόγο να δούμε αν θα μπορέσουν να απαντήσουν ε, τις ερωτήσεις σας. Λέλα Σάντσες. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τερέσα για τις ε, τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε για την έκθεση αυτή, την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική στην ομάδα μας. Θα ήθελα να παραθέσω και τον κύριο Σαραμάκο, βραβείο Νόμπελ ε, λογοτεχνίας που είπε ότι όταν βλέπει κανείς τα πλεονεκτήματα της απελευθέρωσης ε, και τη συγκέντρωση των δύναμης της μεγάλης επιχειρήσης δεκαετία του 1990 είπε ότι η δημοκρατία κινδυνεύει να αποτελέσει ε, ουσιαστικά αντικείμενο κατάχρησης της οικονομικής δύναμης και εμεί είμαστε τη ίδια άποψη. Βλέπουμε ότι έχουν μετατραπεί όλα αυτά σε πολιτικά συστήματα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ε, ε, δεσμούς, να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, να μην ε, παραβιάζεται η κοινωνική δικαιοσύνη ατιμόρυτα. Αν δούμε τις δυνατότητες που δίνονται στους πολίτες ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες ε, απαιτείται συμμετοχή σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν πρέπει να πάψουμε να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές. Η αναπτυξιακή διαδικασία χρειάζεται πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς με σωστό ε, ισορροπημένο και δίκαιο ε, θεσμικό σύστημα που θα βοηθήσει τους ανθρώπους στις χώρες αυτές. Οι πιο σημαντικές εμπορικές ε, και πολιτικές δυνάμεις στον πλανήτη υπογράφουν αυτή τη στιγμή μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες. Βλέπουμε στην Κολομβία, για παράδειγμα, τεράστιο ρυθμό δολοφονιών, στο Μεξικό δολοφονίες δημοσιογράφων, και δολοφονίες ε, χωρικών ε, σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη αναπτύσσοντας ε, πλαίσια τα οποία θα ενισχύουν τα σημερινά συστήματα. Πρέπει να ελέγξουμε τις κρίσιμες δομές στις χώρες αυτές και αυτό θα εξαρτηθεί από την Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις αντιπροσωπείες και θα πρέπει να ε, ε, ορίσουμε σωστού διευθυντέ στο, Ευρωπαϊκό, στο Συμβούλιο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Πρέπει να βρούμε πού βρίσκονται τα κενά, να ενισχύσουμε ε, το προσωπικό και στις αντιπροσωπείες και στα, ευρωπαϊκά, και στα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Και στην Ευρώπη όμως υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χρειάζεται να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για, σε, σε βάρος όσων προβαίνουν σε καταχρήσεις. Υπάρχουν νομικές υποχρώσεις και πρέπει να γίνονται σεβαστές και να αποφύγουμε τα δικά μας θεσμικά όργανα να συμμετέχουν σε οτιδήποτε μπορεί να βλάψει τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να εξετάζεται διαρκώς ποια πράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις, πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις και στο πολιτικό επίπεδο, ώστε να υπερασπιστούμε αυτό το κεκτημένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να σας Αν διαβάζετε από κείμενο, σας παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν οι διερμηνέεις διότι δεν το είχαν από πριν και είναι δύσκολο να αποδώσουν τις λεπτομέρειες. Μαρία εγώ παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσένα Τέρεζα. Περιμένω να βάλεις τα ακουστικά σου. Θα περίμενω, θα περίμενω. Ευχαριστώ και πάλι λέω και εσένα Τερέζα για την πάρα πολύ ε, θετική έκθεση. Η κοινωνία των πολιτών όντω παίζει ρόλο κλειδί και ιδίω όταν πρόκειται για τη φροντίδα των μειονοτήτων, οι ομάδων που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία ε, για τα δικαιώματα των γυναικών, για το περιβάλλον. Για παράδειγμα, η εγκληματικότητα σε βάρος του περιβάλλοντος. Πώς μαθαίνουμε για τα πράγματα αυτά από τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, η οποία η κοινωνία των πολιτών έχει και την δυνατότητα αλλά και το δυναμικό να οδηγήσει και σε μια εξισορρόπηση των συμφερόντων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό συμβαίνει βεβαίω και στι αναπτυσσόμενε χώρε, όπω και εδώ. Όπω είπε και ο προηγούμενο συνάδελφο μου αλλά και ο Σαρλ Γκούρεν. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Έχω να πω και ένα ακόμη, διότι όλα τα άλλα τα είπατε. Χάνουμε και μερίδιο τη αξιοπιστία μα όταν ω Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είναι κάτι προς το δικό μας συμφέρον, είμαστε διατεθειμένοι και διατεθειμένες να συνεργαστούμε με απολυταρχικά καθεστώτα και με δικτάτορες, από την άλλη μεριά όμως δακτυλοδεικτούμε για παραβιάσει ανθρώπων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε συνεπείς και να μην συνεργαζόμεθα με δικτάτορες για δικό μας όφελος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Εσείς ήταν η τελευταία. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακούσατε. Πατρίς Λενορμόν που είσαστε από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα βεβαίως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την ε, σημασία της έκθεσης εφόσον μιλάμε για 100 χώρες έχουν είτε περιορισμούς ε, φυσικούς ε, ή άλλους για το θέμα αυτό. Εδώ και δέκα χρόνια ήταν κυρίω οργανώσει Κοινωνία πολιτών για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που ήταν θύματα τη συρρήκνωση του χώρου. Σήμερα είναι όλες οι ΜΚΟ, ακόμα και αυτέ που εργάζονται για θέματα που δεν είναι ευαίσθητα για τι χώρε εταίρου. Ευχαριστώ και υποστηρίζουμε πλήρως αυτή την έκθεση. Θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε κάθε παράγραφο της έκθεσης αυτής όσο έχει σήμερα και νομίζω ότι αυτό είναι σπάνιο. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό είπε ο κύριος Γκόμες για να υπενθυμίσω ότι το 2012 υιοθετήσαμε ριζική αλλαγή στην προσέγγιση μας στην κοινωνία των πολιτών για να συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε και τις οργανώσεις που είναι οι πρωταγωνιστές ε, της ανάπτυξης επιτόπου αλλά και είναι επίσης οι πρωταγωνιστές της διακυβέρνησης. Έπρεπε λοιπόν να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, τη συμμετοχή της, να ενισχύσουμε τις ικανότητές της και το χώρο της. Έχουμε έναν απολογισμό των όσων έγιναν εδώ και τέσσερα χρόνια. Νομίζω τη στείλαμε την έκθεση αυτή. Δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για τη συμφωνία της ε, Κοτονού. Θα θέλαμε να το κάνουμε και στο φόρουμ του Ιουλίου θα θέλαμε ε, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό εφόσον ε, εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής με την Αφρικανική Ένωση τον Νοέμβριο θα θέλαμε μια πραγματική συζήτηση με την Ένωση αυτή που είναι κάτι αρκετά δύσκολο θα σας καλέσω λοιπόν να έχετε μια συζήτηση μαζί μας εν ώψη αυτούς τους φόρουμ και να εξετάσετε τον απολογισμό. Δεύτερο σημείο της έκθεσης, το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, στην περίοδο του προγραμματισμού του προηγούμενου εργαστήκαμε πολύ για την αρνητική άποψη ε, και θεσπίσαμε πολλούς μηχανισμούς για να υποστηρίξουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΜΚΟ που είχαν πληγεί έναν μηχανισμό υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε ε, ε, περίοδο κρίσης και νομίζω ότι έχουμε ε, πάρα πολλούς κάθε μέρα που κινδυνεύουν να θανατωθούν, να πεθάνουν. Χάρη σε αυτό το κοινοβούλιο και σε αυτό το μηχανισμό μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πρέπει να διατηρήσουμε τον μηχανισμό για να μην υπάρχει η ίδια κατάσταση στο μέλλον. Στα πλαίσια της συζήτησης για τον προγραμματισμό θα πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μερικοί άλλοι όπως οι Νορβηγοί φίλοι μας ασχολούνται με το θέμα αυτό. Ένα δεύτερο σημείο όπου δεν κάναμε αρκετά πράγματα και πτονίζεται στην έκθεση είναι ότι να εργαστούμε λιγότερο, με λιγότερο αμυντικό τρόπο για να υποστηρίξουμε τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στην κοινωνία των πολιτών σε ορισμένε χώρε, τι δράσει τη κοινωνία των πολιτών που εργάστηκαν για νέου χώρου, για νέου νόμου που άνοιξαν πόρτε και αυτό ε, θα γίνει στα πλαίσια της του μελλοντικού προγραμματισμού. Μην μιλάμε μόνο για τα αρνητικά θέματα θα πρέπει να μιλάμε ε, και με τρόπο πιο θετικό και πιο επιθετικό για τις καλές πρακτικές. Στο νακτή του ελεφαντοστού υπάρχουν δράσεις θετικές, πρέπει να τις υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουμε τις οργανώσεις που ε, τις υλοποιούν και όταν συζητήσουμε το Κοινοβούλιο θα έχουμε προτάσεις για να ε, συνεχίσουμε ε, να περιορίζουμε τα προβλήματα, να προστατεύουμε ε, τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και παράλληλα αυτό που τονίζεται στην έκθεση με το θεματικό μέσο για την κοινωνία των πολιτών να υποστηρίξουμε καλύτερα στο πλαίσιο το θετικό την κατάσταση και να μην είμαστε μόνο ε, αμυντικοί, αλλά να είμαστε και επιθετικοί. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την καλή έκθεση που έρχεται ε, σε καλή στιγμή, διότι υπάρχουν πολλά θέματα για την κατάσταση. Πολλές ΜΚΟ δεν μιλάνε μόνο για τη συρρήκνωση του χώρου, αλλά και για την εξάλληψη του χώρου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ήθελε και κάποιος άλλος να μιλήσει. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ναι, παρακαλώ κύριε Ρώσο, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την πολύ επίκαιρη έκθεση αυτή. Ήθελα και εγώ να τονίσω πόσο σημαντική είναι η συρρήκνωση του χώρου Τη κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρε. Εμεί έχουμε σαφή ε, πολιτική δέσμευση ω εντολή τη κυρία Μογκερίνη και των κρατών μελών. Το νέο σχέδιο δράση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα για το περίοδο 2015-2019 που υιοθετήθηκε από τους Υπουργούς τον Ιούλιο του 2015 αναφέρει τη δέσμευση ε, για την ενίσχυση και τη χειραφέτηση της κοινωνίας των πολιτών. Στο σχέδιο δράσης ε, αναφέρεται η ανάληψη δράσης ε, αναφέροντας και, τις, ε, και τους περιορισμούς ε, του δικαιώματος συνεταιρίζεστε και συνέρχεστε. Τα ζητήματα αυτά έχουν συζητηθεί σε διμερείς συνεδριές, σε πολυμερείς συνεδριές και σε διεθνή φόρα, όπως και στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των ΗΠΑ. Εθνών. Το σχέδιο δράσης επίσης περιλαμβάνει μία δέσμευση προληπτικής δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, εντοπίζοντα τι απειλέ αυτέ και λαμβάνοντα μέτρα για την αντιμετώπιση τους αρκετά νωρί. Πρέπει να δράμε πιο γρήγορα, αποθαρρύνοντα κυβερνήσει και κοινοβούλια από την υιοθέτηση τέτοιων μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει προσπάθειε ε, για να γίνει η δουλειά τη πιο συνεκτική στο πλαίσιο τη δημοκρατία, τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη κοινωνία των πολιτών. Έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή τη, ένα ευρύ διπλωματικό δίκτυο, νέε αντιπροσωπείε ε, και πρεσβείε κρατών μελών και το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα του κόσμου με σημαντικό προϋπολογισμό για τα ανεπτυξιακά έργα. Απαιτείται στενό συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, άλλων υπηρεσιών τη Κομισιόν, των κρατών μελών και μεταξύ των ε, κεντρικών γραφείων και των αποστολών. Το νέο σχέδιο δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία αναγνωρίζει ότι η σοβαρότητα του προβλήματο ε, τη ρύθμιση του χώρου απαιτεί συνεκτική και αποτελεσματική απόκριση με διπλωματική δράση, συντονισμένες ε, διπλωματικές πολυμερείς προσπάθειες και ε, συντονισμό με τους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποφυλάκηση ε, κρατουμένων δημοσιογράφων κτλ. και ακτιβιστών που έχουν φυλακιστεί λόγω της δράσης τους ε, για την υπερασπιστή των ανθρώπινων δικαιωμάτων συζητώνται τακτικά ε, σε διάφορου συμβατισμούς του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τερέσα, θέλατε να μα ε, πείτε κάποια συμπεράσματα. Ναι, ευχαριστώ πολύ Λίντα. Ευχαριστώ όλες και όλους για τα σχόλιά σας. Θα τα σημειώσω, τα λαμβάνω υπόψη. Έχουμε κάποιο χρόνο ακόμη για να ε, δούμε και τις ε, τροπολογίες. Βεβαίως και συμφωνώ ότι πρόκειται και για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εδώ στην ίδια την Ευρώπη και ότι εμείς πρώτες και πρώτοι θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα πριν να μιλούμε σε άλλες χώρες για δημοκρατία. Οι συναδέλφισέ μου και οι συναδελφοί μου μίλησαν για ορισμένε άλλε χώρε, όπω για την Ουγγαρία. Και μάλιστα και προ λίγων εβδομάδων ψηφίστηκε ένα ψήφισμα. Δεν μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί κανείς ότι δακτυλοδεικτούμε τους άλλους και ότι αποστρέφουμε το πρόσωπό μας από ε, πράγματα που συμβαίνουν εδώ παροιμήν. Όταν μιλούμε στην έκθεσή μου για αναπτυσσόμενες χώρες, δεν σημαίνει αυτό ότι παραμελούμε την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναφέρω ονομαστικά χώρες μέλη της Ένωσης, διότι συζητήσαμε στην Υποεπιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και ήθελα να συζητήσουμε και εδώ, στην Επιτροπή ΔΕΒΕ, που ούτως ή άλλως το αντικείμενό μας είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι είναι σωστό άλλωστε να σημειώνει κανείς ακόμα και τις ε, μικρές επιτυχίες εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Αυτό που συνέβη για παράδειγμα πρόσφατα στο Μεξικό αλλά και όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Νομίζω ότι χωρίς να κάνουμε προσπάθεια να καταδικάσουμε πολιτικά ρεύματα, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τονίζονται. ερχόμενοι σε επαφή με τους πρέσβεις των χωρών αυτών, μπορούμε να τους θέσουμε τα θέματα υπόψη και νομίζω ότι είναι σωστό να τονίσουμε και παραδείγματα όπου υπάρχει μια συνεργασία και μια αμοιβαία προσέγγιση. Πρέπει να τονίζονται και αυτά. Ώστε να ξεφύγουμε από τα πλαίσια της αντιπαράθεσης και της εχθρικής διάθεσης. Εκεί βλέπω να βρίσκεται ο ρόλος μας, ένας ρόλος διαμεσολαβητού. Και είναι σημαντικό βέβαια να συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ακόμη να φροντίσουμε να θέσουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας την προστασία των ακτιβιστών και ακτιβιστριών. Αυτό πρέπει να εκφραστεί με απόλυτη σαφήνεια, διότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, διότι συχνά διακινδυνεύει και η ζωή του. Ευχαριστώ με Τερέσα. Να υπενθυμίσω 20, 21η Μαΐου, 10 η ώρα το πρωί, ε, ε, ε είναι 21η συγγνώμη Μαΐου. Είναι η προθεσμία για υποβολή τρομολογιών. Πάμε στο σημείο 6. Απόδοση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών στην παροχή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε κάποιου ομιλητέ που μπαίνουν στην αίθουσα τώρα. Έχουμε να συζητήσουμε ένα σημαντικό θέμα τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Τίθε το θέμα του πώ τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη αντιμετωπίζουν το ζήτημα τη ε, παροχή ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και τι αποτελέσματα φέρνει η Κομισιόν ε, όσον αφορά την αναζήτηση ευθυνών και λογοδοσία από τα κράτη-μέλη. Όπω ξέρετε, το 2005 ε, υποχρεώθηκαν τα κράτη-μέλη για παροχή αναπτυξιακής βοήθεια 1,7% του ΑΕΠ του. Ε, στο μεταξύ, ε, αργότερα τα κράτη-μέλη ανέφεραν την οικονομική κρίση για τη μη επιτεύξη αυτού του ποσοστού. Ο ΣΑ εκπονεί μια έκθεση ετησίω για τις αποδόσεις των κρατών μελών. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Χαζιασούτε που είναι επικεφαλής ε, της γραμματείας του ΩΣΑ για θέματα οικονομικά και την κυρία Μελό που είναι ε, αναπληρωτής νεματάρχης της Γενικής Διεθνής ΔΕΒΚΟ. Θα μας μιλήσουν για τα τελευταία νούμερα. Έγινε μια συζήτηση και στο Συμβούλιο ε, Υπουργών Ανάπτυξη στις 19 Μαΐου όπου αυτό συζητήθηκε από τους υπουργού εκεί και τέθηκε και άλλο ένα ζήτημα που θα συζητήσουμε αργότερα σήμερα θα ψηφίσουμε τη συνένεση για την ανάπτυξη. Κάτι πρέπει σημαντικό για τη δεσμεύση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπλήρωση των ε, στόχων βιωσιμής ανάπτυξης μέχρι το 2030. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα σα στείλουμε και ένα αντίγραφο του ε, δελτίου τύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Απριλίου που αναφέρει τι επιδόσει ε, των κρατών μελών. Πέντε κράτη-μέλη από τα 28 τα οποία έχουν επιτύχει τώρα το στόχο του 1,7%. Υπάρχει μικρότερος στόχος για τις νέες 12 χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγιναν μέλη μετά το 2004. Είναι χαμηλότερος ο στόχος για αυτές. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν δίνω το λόγο πρώτα στον κύριο Σούτε. Να μας πείτε λοιπόν ε, πώς βλέπετε τα πράγματα από την πλευρά του ΩΣΑ και πώς, ε, ποια είναι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Έχετε το λόγο κύριε Σούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας ξανακαλείτε φέτος uh, τον ΩΣΑ να σας δώσουμε μια γενική εικόνα όλων uh, των αριθμών. Να, θα καλύψω τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, θα σας παρουσιάσω την προσέγγιση μας uh, για τα ODA και πώς τηρούμε τις δεσμεύσεις και των κρατομελών αλλά και της διεθνούς κοινότητας και μετά θα επικεντρωθώ στα άλλα νούμερα και τέλος θα μιλήσω για τις εσωτερικές μεταναστευτικές ροές υπήρξε σημαντική αλλαγή ε, αλλαγή, μεταβολή Λοιπόν, Όσοι γνωρίζουν ε, τα νούμερα ODA και τον τρόπο συλλογής τους, θα σας πω ότι τα νούμερα που θα σας παρουσιάσω είναι τα προκαταρκτικά νούμερα. Είναι αυτά που αναφέρουν τα κράτη-μέλη, δηλώνουν στον ΩΣΑ. Και μετά, ε, με προθεσμία, η προθεσμία αυτή είναι οι αρχές Απριλίου και στη συνέχεια μας στέλνουν και πολλά νούμερα σε επίπεδο δραστηριοτήτων. Αυτά τα στοιχεία δραστηριοτήτων αφορούν την διασφαλίση και στη συνέχεια δημοσιεύουμε τα νούμερα επίπεδου δραστηριότητας το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Αυτό θα μπορέσετε να δείτε αν θέλετε να περάσετε ένα συναρπαστικό κυριακάτικο απόγευμα, μπορείτε να πάτε στο ECD DAC Development Finance, όπου θα βρείτε στη σελίδα μας αυτή, όπου θα βρείτε όλα τα νούμερα, ε, πάρα πολλά έργα, χιλιάδες έργα, τα οποία ε, δηλώνονται σε εμά και εκεί θα βρείτε πρόσβαση στα δεδομένα. Ε, και από πολλές οπτικές γωνίες και με πολλές διαφάνειες και εικόνες που σας δίνουν, πιστεύω, μια πολύ σαφή εικόνα του πώς ε, αναπτυστεί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και πώς στηρείται από τα κράτη-μέλη. Θα ξεκινήσω λέγοντας με την πρώτη μου διαφάνεια ότι προφανώς όπως γνωρίζουμε όλοι η ατζέντα δράσεων ε, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας μας παρέχει ένα πολύ φιλόδοξο πλαίσιο το 2015 τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ένα πολύ φιλόδοξο βασικό σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και για την τήρηση της Συμφωνίας των Παρισιών του ίδιου έτους. Και αυτό μας οδήγησε να σκεφτούμε στον ΩΣΑ, αλλά και στην Επιτροπή ε, Αναπτυξιακής Αρρωγής. Ε, μας έκανε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη χρηματοδοτική πρόκληση. Οι προσπάθειες μας ε, βασίζονται σε, τρία, σε τρεις τομείς. Ε, στην μέτρηση, όπου θα εστιαστώ και σήμερα, στην υπαρχή κινήτρων και την κινητοποίηση είναι ο δεύτερος πυλώνας και η εκμάθηση είναι ο τρίτος ε, πυλώνας. Εκμάθηση και δημιουργία εταιρική σχέση. Αυτό είναι η πολιτική πτυχή του έργου μας. Ό,τι και να κάνουμε, αυτό πρέπει να γίνεται σε στενή συνεργασία με άλλες χώρες, με τα ΗΕ, με τον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζει το σημαντικό ε, συμμετέχον στο πλαίσιο τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και η κοινωνία των πολιτών φυσικά, αλλά και οι πιο σημαντικοί συμμετέχοντες είναι οι χώρες, οι χώρες αποδέκτες της βοήθειας. Δείχνω αυτή τη διαφάνεια διότι γνωρίζω ότι πολλά από αυτά τα σημεία που θα έχετε καλύψει εδώ στη συζήτηση, να πω ότι στην πάνω δεξιά πλευρά Βλέπετε ζητήματα όπως ο εξυγχρονισμός της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και κάτι άλλο στο οποίο θα αναφερθώ σήμερα. Ε, εστιαζόμαστε και σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες που παίρνουν από ένα πολυμερές σύστημα. Ε, έχουμε και τους παρόχους Νότου-Νότου και το TOSSD. SSD. Ε, όλο και περισσότερη βοήθεια παρέχεται από ε, φορείς ε, στο Νότο. Και μετά έχουμε το 2-SSD που είναι ένα σύστημα μέτρησης το οποίο μπορούμε να καταγράψουμε τις ροές από το βορρά προς τον νότο και πιο ευρέως ε, πέραν της επίσημης αναπτυξικής βοήθειας. Είναι σημαντικός τρόπος ε, που θα μας βοηθήσει στο μέλλον να μετράμε κατά πόσο ο Βορράς ε, πληρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όσον αφορά την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Στο, με μπλε χρώμα στα αριστερά βλέπετε τα εργαλεία του ιδιωτικού τομέα, κάτι, ένα έργο που συνεχίζεται σήμερα. Προσπαθούμε να καταγράψουμε το έργο των ε, χρηματο, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση της ανάπτυξης στη Γερμανία, στις κατοχώρες, ε, στη Σουηδία και βρισκόμαστε εν μέσω της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό. Δηλαδή σε ποιο βαθμό θα λαμβάνονται υπόψη την επίσημη αναπτυξική βοήθεια όλες αυτές οι δράσεις. Τώρα η κινητοποίηση διαφορετικών ε, πόρων είναι ένα σημαντικό θέμα για την επίσημη αναπτυξική βοήθεια, η οποία είναι πολύ σημαντική για τις χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικές ανάγκες. Πάντα τίθεται λοιπόν το θέμα της ισορρόπησης ε, μεταξύ έξυπνης χρήσης της ε, επίσημης αναπτυξικής βοήθειας και διασφάλισης της διάθεσης της χρηματοδότησης ε, για τις χώρες που τη χρειάζονται περισσότερο. Όσο μεγαλώνουμε την πίτα ουσιαστικά, όσο περισσότεροι πόροι υπάρχουν διαθέσιμοι, ε, τόσο περισσότερα χρήματα υπάρχουν για αυτές τις χώρες ε, που έχουν μεγάλες ανάγκες. Για την κλιματική χρηματοδότηση δεν έχω να πω κάτι άλλο και για τη μεικτή χρηματοδότηση ουσιαστικά είναι συνεργασία μεταξύ ε, δημόσιας ε, και ε, ιδιωτικής χρηματοδότησης. Θέλουμε να καταλήξουμε να δημιουργήσουμε και κάποιες αρχές και γραμμές πολιτικής για τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτών. Και μετά με MOV κάτω δεξιά βλέπουμε διάφορες προσπάθειε σε θέματα πολιτική για την εκμάθηση. Πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο αποτελεσματικέ εταιρικέ σχέσει, κινητοποιώντα την αναπτυξιακή χρηματοδότηση ε, σε τεχνολογικά θέματα. Ένα συναρπαστικό τρόπο συνεργασία σε δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κάτι που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το μέλλον. Ε, κάτι που θα κρατήσει δεσμευμένου όλου ε, με την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Και μετά έχουμε ένα εμβληματικό έργο προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι σημαντική η δημόσια και η ε, ιδιωτική χρηματοδότηση αλλά και οι φιλανθρωπικές ε, δράσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να διερευνήσουμε όλες αυτές τις αλληλεσυνδέσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών χρηματοδοτικών ε, ροών ώστε να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους. Θα ήθελα να εστιαστώ τώρα λοιπόν περισσότερο στους αριθμούς και να σας δώσω μια εικόνα των νούμερων για το 2016. Τι βλέπουμε εδώ. Με την μπλε γραμμή, στην μπλε γραμμή βλέπετε ότι η επίσημη αναπτυξική βοήθεια έχει αυξηθεί το 2016 ουσιαστικά έχουμε μια πρωτόγνωρη ε, υψηλή τιμή έφτασε τα 142,6 δισεκατομμύρια δολάρια η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πρόκειται για τεράστια αύξηση. Ε, είναι πολύ σημαντική αν λάβει κανείς υπόψη την αύξηση του 8,9% και κοιτώντας την κόκκινη την κόκκινη γραμμή βλέπετε ε, την αναλογία μεταξύ επισήμης αναπτυξιακής βοήθειας και ΑΕΠ και αν συγκρίνεται μεταξύ 2015 και 2016 παρατηρείται αύξηση σήμερα 3,2% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Um, this Έτσι αποκτάτε μια εικόνα του, σε εξέλιξη της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας από το 2000 και μετά. Με μπλε χρώμα έχετε τη διμερή βοήθεια, με γαλάζιο την πολυμερή επίσημη ανάπτυξη βοήθεια, με κόκκινο την ανθρωπιστική βοήθεια, με πράσινο που αυξάνεται σημαντικά είναι τα κόστη των χρηματοδοτών για τους μετανάστες. Το αναφέρουμε και πριν, θα επανέλθω σε αυτό αργότερα και με ΜΟΒ έχουμε την ανακοψη χρέους. Οπότε έχω να πω ότι ουσιαστικά η διεθνή κοινότητα και τα μέλη εδώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διπλασιάσει σε σχέση με το 2000 την βοήθεια. Είναι κάτι για το οποίο όλοι πιστεύω είμαστε περήφανοι. Το 2016 σημαντική παραγωγή ήταν η αύξηση αφενός ε, του κόστους για τους ε, πρόσφυγες και αφετέρου το κόστος ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό βλέπετε εδώ με το κόκκινο και το πράσινο χρώμα. Παρ' όλα αυτά πρέπει όμως να πούμε ότι ουσιαστικά αν αφαιρέσουμε την αύξηση του internal Refugee Cost, εξακολουθούμε να έχουμε αύξηση της επίσημης ε, αναπτυξιακής βοήθειας ε, κατά 7,1% με το προηγούμενο έτος ε, σε πραγματικά νούμερα. Να σας πω Δύο λόγια για το Internal Refugee Cost και την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, ε, είναι η κόκκινη περιοχή που βλέπετε εδώ, που έχει αναπτυχθεί πολύ σημαντικά από το 2014 και μετά. Αυτό το κόστος έχει αυξηθεί κατά 28% σε πραγματικά νούμερα σε σχέση με το περασμένο έτος σε 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής από 12,1 δισεκατομμύρια το προηγούμενο έτος και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ουσιαστικά 10% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας ε, χρησιμοποιήθηκε υψηλότερο ποσοστό από πέρυσι που είχαμε ήδη το υψηλότερο ποσοστό του 9,2% και έχουμε πολλές χώρες όπου αυτά τα κόστη, τα internal refugee costs αντιστοιχούν στο 10% της ε, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Μιλάμε για 11 μέλη ε, της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας και επίσης τέσσερις χώρες ε, έχουν τέτοια δαπάνη σε του 20%. Το 2016 τόσο η ανθρωπιστική βοήθεια και το Internal Refugee Cost αντιστοιχούν σε ε, ή αρκετά υψηλό ποσοστό του συνολικού ε, της ελληνικής επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Υπάρχουν και κάποιοι τομείς ε, που θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν πιο στενά από τα μέλη της Αναπτυξιακής Επιτροπής είναι ότι η αρκετα υψηλο ποσοστο του συνολικου τη ελληνικης επισημης αναπτυξιακης βοηθειας υπαρχουν και καποιοι τομεί που έχει απο τα μελη της αναπτυξιακή επιτροπης ειναι από το 2014 μέχρι το 2016 τόσο για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αλλά και για την Αφρική για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, υπήρξε πτώση του 3,9% σε 24 δις ε, το 2016 και για την Αφρική αν δούμε την υποσαχάρη Αφρική για παράδειγμα η πτώση ήταν 0,7% σε σχέση με το 2015 σε 24 δηλαδή δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής είναι λοιπόν συγκεχημένη. Η εικόνα είναι μεικτή. Έχουμε διαφορετικά σενάρια σε διαφορετικά μέρη. Για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια γενικώ τα στοιχεία μα αφήνουν ικανοποιημένου, αλλά έχουμε και αύξηση του κόστου internal refugee, αύξηση τη ανθρωπιστική βοήθεια και πτώση τη βοήθεια προ την Αφρική και τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Και αυτό φυσικά είναι κάτι που είχε συμφωνήσει η Διεθνή κοινότητα να αυξήσει. Γενικά λοιπόν οι επιδόσεις μας δεν ευθυγραμμίζονται με τις δεσμεύσεις. Οπότε θα πρέπει να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στα νούμερα που μας αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τη δυναμική γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης της ανθρωπιστικής βοήθειας της αύξησης της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, κατευθύνεται στη Συρία και στις γειτονικές χώρες πιθανότατα τα τέλη του έτους λοιπόν όταν θα ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στα στάσεις αυτές θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Όπως βλέπουμε τις ε, διμερείς επιδόσεις ε, δωρητών, βλέπουμε σε δολάρια. Ε, στην αριστερή πλευρά βλέπω ότι οι μεγαλύτεροι δωρητέ και θα μας εκπλήσει είναι οι ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Ιαπωνία και Γαλλία. Παρατηρείται ότι υπάρχει αυξή σε 22 χώρες ε, σε μερικές περιπτώσεις αυτό οφείλεται στις ε, προσφύγες ε, στις δωρήτρες χώρες κάποιες χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάποιες περιπτώσεις απλά υπάρχει διαφορετικός τρόπος αντιμετώπιση των προσφύγων στις δωρήτρες χώρες οι 20 ε, χώρες DAC που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί συνολικά το ύψος του σε επίσημες αναπτυξιακές βοήθειες ήταν 81,3 ε, δισεκατομμύρια, δηλαδή με αύξηση 13,1%. Και σε σύγκριση με το συνολικό τους ΑΕΠ είναι 0,51% η αναλογία αυτή. Εδώ βλέπετε λοιπόν τώρα την σύγκριση με το στόχο του 7% των Ηνωμένων Εθνών ε, για ε, το 0,7% σε σχέση με το ΕΠ. Έχετε εδώ Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Δανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο που κατάφεραν να επιτύχουν αυτό το 0,7% πέρυσι. και κάτω δεξιά, στη δεξιά πλευρά του βλέπετε ότι η αναλογία για κάποια μέλη ήταν μηδεν ε, κάτω από μηδέν. Ήταν τα χαμηλή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που συμμετείχαν στον ΤΑΚ ε, παρήχαν 1,12% του ΑΕΠ και 2% Τώρα κάποιοι σημαντικούς πόρους παρότι ότι δεν είναι μέλη του ΝΤΑΚ για την επίσημη ανάπτυξη βοήθεια. Έχω ακόμα τέσσερις διαφάνειες, κυρία Πρόεδρε. Ε, τελειώνει ο χρόνος, λέει ο Πρόεδρος, ε, και χρειαζόμαστε να ακούσουμε και την Κομισιόν. Ε, θα ήθελα να σας πω λοιπόν ένα βασικό ζήματα, ζήτημα ήταν το κόστος ε, των προσφύγων στις δωρετές χώρες. Ε, ορίστηκε για το δεκαετία του 80 και κατέστησε σαφές ότι οι κανόνες που υπήρχαν δεν ήταν επικαιροποιημένοι. Η διαδικασία ουσιαστικά συνεχίζεται για τη διευκρίνηση των κανόνων αυτών. Έχουμε μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με το θέμα αυτό η οποία ουσιαστικά όπως ανακαλύψαμε και μέσω μιας, ε, όπως, μέσω μιας έρευνας ε, ανακαλύψε ότι πρέπει να εστιάσει το έργο της ε, στους εξής τομείς. και όταν υπάρχουν διαφορές στις πρακτικές αυτές αφορούν τις κατηγορίες των προσφύγων, του δεσάσυλο, πρόσφυγες, τι τύποι δαπανών καλύπτονται, προσωρινή διαβίωση, διοικητικά κόστη, καθώς και μεθοδολογίες που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κόστους. Και στην τελευταία διαφάνεια βλέπετε ότι εδώ απαιτούνται πέντε διευκρινήσεις. Ποια είναι η λογική για την συμπερίληψη του κόστους για πρόσφυγες στις δωρήτε χώρες στην επισημένα αναπτυξιακή βοήθεια. Ποιέ κατηγορίες προσφύγων είναι επιλέξιμες για να συμπεριληφθούν τίθεται το ζήτημα του ότι το κόστος μόνο των πρώτων 12 μηνών πρέπει να καλύπτεται οπότε τίθεται το ερώτημα του πότε αρχίζουμε να μετράμε και πρέπει μετά να δούμε πώς θα κατανοήσουμε τα διάφορα, να συνεννοηθούμε ποια θα είναι τα στοιχεία κόστους που θα συμπεριλαμβάνονται και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους. Στόχος μας είναι εντάξει, να υιοθετήσει τις ευκρινήσεις αυτές τον Ιούλιο στην ε, Σύνοδο Κορυφή υψηλού επίπεδου, δηλαδή των Υπουργών των Μελών τη ΔΑΚ για επικύρωση του Οκτώβριου του 2017. Οπότε, όχι μόνο λόγω των προσφύγων που έρχονται στην Ευρώπη, αλλά και λόγω της συντηρητική αυτής διευκρίνησης θεωρούμε ότι θα έχουμε σημαντική μείωση του κόστους ε, για τους πρόσφυγες στις δωρήτρες χώρες. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ για την σε βάθος ανάλυση των τεκτενομένων για το κόστος των προσφύγων στις ίδιες τις δωρήτρες χώρες. Θα σας παρακαλέσω σας κυρία μου να μας πείτε τι σημαίνουν αυτά. Αλλά βέβαια όχι, μη, μακρηγορήσετε τόσο πολύ. Η κυρία Μερελό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα Ηνωμένα ΕΕ χώρες χώρε μέλη αποτελούν ε, σημαντικού συνεισφορεί στην θετική αυτή εικόνα που παρουσίασε προηγουμένω ο συνάδελφό μου. Συνολικά, μιλούμε σε ευρώ πλέον, έτσι, όχι σε δολάρια, άρα υπάρχει κάποια διαφορά, έτσι δεν είναι. Οι χώρες μέλη της Ένωσης έδωσαν 75,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2016. Αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2015. 2015. Και πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά έτος που αυξάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνειφορά της. Άρα είναι πράγματι θετική εικόνα. Οι χώρες μέλη εκπροσωπούν το 58% συνολικά της ODA, της επίσημης δηλαδή ε, ε, στήριξης για την ανάπτυξη. Πέντε χώρες μέλη έχουν φτάσει το 0,7%. Επανεπιβεβαιώθηκε τον Μάιο του 2015 από όλες τις χώρες μέλη. Ο στόχος αυτός. Οι περισσότερες χώρες μέλη αύξησαν τις παροχές στην ODA και μόνο πέντε τη μείωσαν το 2016 σε σύγκριση με το 2015. Αν εξετάσουμε τώρα την πρόοδο που κάνουμε προς την ε, στο συλλογικό στόχο το 0,7% του ΑΕΠ, για το 2016 επιτύχαμε 0,51% που είναι και το υψηλότερο ποσοστό μέχρι τώρα. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει ακόμα τον τελικό στόχο, αλλά είναι σημαντική η πρόοδος και υπογραμμίζω ότι αν εξετάσουμε και τους υπόλοιπους δωρητές, η αναλογία τους σε σχέση με το ε, ΑΕΠ είναι μόνο 0,21%. Αν εξετάσουμε τώρα περισσότερο το κόστος για τους πρόσφυγες στι δωρήτριε χώρε που προσφεύγουν στι δηλαδή στις χώρε, χώρες, έχει αυξηθεί και αυτό τα τελευταία τρία χρόνια. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι στι χώρες μέλη τη Ένωσης αυτές μπόρεσαν να αυξήσουν την ODA και καθαρά και στα κόστη των in-donor refugees. Και αυτό είναι σημαντικό. Στο σύνολο η αύξηση της ODA ήταν 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά η αύξηση για το κόστος των Ιντόνων ήταν 1,9 δισεκατομμύριο, δηλαδή 25% της συνολικής αύξησης. Χαμηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια, το 2015, η αύξηση για το κόστος των Ιντόνων ήταν 64% της συνολικής αύξησης, ενώ το 2014 ήταν 56% της συνολικής αύξησης της ODA, της επίσημης δηλαδή αναπτυξιακής ε, στήριξης. Άρα βλέπουμε μία μείωση. Κατά ένα τέταρτο περίπου συνολικά. Αυτό βέβαια οφείλουμε να το σημειώσουμε. Το τελευταίο που θέλω να σας ε, θέσω υπόψη, ότι έχουμε ακόμα μια ανησυχία για τη στήριξη προς αναπτυσσόμενες χώρες. Ακόμα δεν έχουμε νούμερα δυστυχώς, διότι δεν έχουμε επαρκείς λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να κάνουμε ανακετά ανάγλυφα δηλαδή τα δεδομένα για να μπορέσουμε να τα ε, συμπήξουμε σε... Έχουμε ένα της τάξης του 0,11% της ODA για τις ελάχιστα αναπτυσσόμενες χώρες που είναι και πολύ χαμηλότερο στο ενδιάμεσο διάστημα με 0,15% και πηγαίνει για το 0,20%. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι ε, ε, βλέπουμε μια τάση η οποία αυξάνεται. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθούν οι χώρε μέλη για να κάνουν κάποια πρόοδο εν προκειμένου. Θα σταματήσω εδώ και σα ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, σα ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο, γιατί ήσασταν πολύ ακριβεί και πολύ σύντομοι. Τώρα, ορισμένοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ να αυτοπεριοριστείτε σε ένα χρονικό όριο των δύο λεπτών για να μπορούμε, προλάβουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Does Εκτός από τα ονόματα που ανέφερα άλλους κανείς. Σαρτζεντίνη. Άρα, το πολύ δύο λεπτά είναι κάθε μία και ο καθένας από εσάς. Τερέσα Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πάρα πολύ σύντομα. Έχω μια ερώτηση. Όταν μιλάτε ε, για τα δαπάνε ε, των προσφύγων, ποιοι λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια ακριβώς ε, μίλησα για το Λίβανο προηγουμένως. Στο Λίβανο, ε, στην κοιλάδα της Μπεκά, όπου υπάρχουν πάνω από 2.000 κέντρα προσφύγων. Ε, με, έχουμε καταβλισμούς, καμιά δεκαριά καταβλισμούς στο καθένα όπου ζουν 20-30 οικογένειες βλέπαμε το σήμα των Ηνωμένων Εθνών, την αποστολή, αλλά δεν ακούσαμε να γίνεται λόγος ε, για τα κονδύλια που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για τη δική μας πρόταση, για τη δική μας συμβολή δεν γινόταν κανένας λόγος. Υπήρχε μόνο το σήμα των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως, ε, ε, έχουμε ε, σημαντική συνεισφορά. Πώς κατανέμονται τα χρήματα, τα κονδύλια. Γιατί να μην ε, αναφερόμαστε πουθενά, να μην φαινόμαστε πουθενά. Γιατί ποιοι λαμβάνουν τα κονδύλια αυτά, οι κυβερνήσεις, η ΜΚΟ. Θα ήθελα επίσης να μάθω εάν η βοήθεια που λαμβάνουν αυτοί οι ε, πρόσφυγες είναι αυτοί μόνο ή έχουν κάποια άλλη βοήθεια. Θα έχουμε τις, ερω... τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Αμιλίτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκθεσή σας. Θα αναφερθώ κυρίως στην κατάσταση ε, των in-donor refugee costs. Μια ερώτηση που ίσως είναι περίπλοκη. Πόσα ε, πώς γίνονται ε, δεκτή, δεκτά, δεκτές αυτές οι δαπάνες, διότι είναι μια πρόκληση και για το μέλλον και αυτό ε, δεν ανήκει στην σφαίρα της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν ξέρω πώς γίνεται η διαπραγμάτευση με τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ, Σαρβόη. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το άρθρο 8 Τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, διευκρινίζει ότι οι εθνικές πολιτικές των κρατών μελών και η αναπτυξική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλληλοενισχύονται. Ε, είναι, γίνεται λόγος για την εκρίζωση της πτώχειας ως βασικός στόχος αυτής της πολιτικής και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τηρούν, τηρούν, σέβονται τους στόχους που έχουν εγκρίνει στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών ή με τις ε, ε, διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και θα ήθελα ε, να αναφερθώ μόνο στις δεσμεύσεις που έχουν αριθμούς ποσοτικούς 0,7% σε σχέση με τον ΑΕΠ ως το 2030. 2005 είχαμε τον είδο στόχο, αλλά το 2015 15 επίση τον ίδιο στόχο, αλλά δεν λειτουργήσε. Αν δεν αλλάξουμε μέθοδο, θα έχουμε την ίδια διαπίστωση το 2030. Το σύστημα δεν θα λειτουργήσει. Ευχαριστώ τον ΩΣΑ και την Κομισιό που μας έδωσαν αριθμούς, στοιχεία, αλλά είναι μια αξιολόγηση εξπόστε με αυτό που με ενδιαφέρει, είναι η προοπτική τι πρέπει να κάνουμε για να επιτύχουμε το στόχο το 2030. Δεν το πράξαμε μέχρι τώρα. Εμείς παρακολουθούμε τα γεγονότα. Αυτό μπορεί να γίνει και από έναν δημοσιογράφο που, ε, που καταρτίζει ένα φάκελο για το θέμα αυτό ή έναν, ε, ε, την, έναν φοιτητή που κάνει την διδακτορική του εργασία. λαμβάνουμε τα στοιχεία με πάρα πολύ καθυστέρηση. Δεύτερον, δεν υπάρχει τίποτα για το μέλλον. Υπάρχουν οι δεσμεύσεις ε, αυτό είναι φιλολογία, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αυτοί που λαμβάνουν τις πληροφορίες είναι παντού στον κόσμο. Ε, ε, μπρος στον ΩΣΑ έρχονται οι χώρες και δίνουν τα στοιχεία τους. Οι αξιολογήσεις ορισμένων κρατών μελών που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και για το μέλλον. Πολύ καλό αυτό, αλλά γιατί αυτά τα στοιχεία δεν κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί τα κράτη-μέλη ενώπιον ε, του ΟΣΑ, των ε, πρεσβευτών ε, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας δίνουν αυτά τα στοιχεία, βιάζονται να δώσουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δικαίωμα να παρακολουθεί αυτή την πολιτική, δικαίωμα να δίνει πολιτική όθηση. Νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε μπρος σε μία μεθοδολογική αποτυχία. Μία μέθοδος η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο την αξιολόγηση ex post και όχι το μέλλον. Πώς μεταφράζονται οι δεσμεύσεις αυτές ε, σε ανάληψη υποχρεώσεων δημοσιονομικών, γιατί κάθε χρόνο ε, δίνονται στοιχεία ε, στην ε, μονάδα την δημοσιονομική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, γιατί δεν υπάρχει δίπλα η αναφορά για τα κονδύλια αυτά για την αναπτυξιακή βοήθεια, για την επόμενη χρήση και τις τρεις επόμενες χρήσεις. Οι χώρες αυτές δίνουν τα στοιχεία στον ΩΣΑ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και βλέπουμε τα στοιχεία, ε, πώς εξελίσσονται. Και γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, αυτό έχει μια σημασία που είναι πάρα πολύ πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, θα είναι ο πρώτος χορηγός, ο πρώτος δωρητής μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, τα 18 δισεκατομμύρια που ξοδεύει το Ηνωμένο Βασίλειο για την επίσημη αναπταξική βοήθεια θα καλυφθούν αυτά τα 18 δισεκατομμύρια. Αν δείτε τα στοιχεία που έχουμε σήμερα τα γνωστά, θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι αν όλα τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει πριν από την αναχώρηση της αντιπροσωπείας μας για την Αντίσα θα μπορούσαμε σε μερικά χρόνια να αντισταθμίσουμε το ποσό που θα μας στερήσει η έξοδος ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μπορεί, ίσως μακρηγόρησα, μπορεί βεβαίως κανείς σε δύο λεπτά να μην πει τίποτα το σημαντικό, αλλά αν δεν κατορθώσουμε να είμαστε σαφείς πάνω στο θέμα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το καθήκον μας, αν είμαστε ε, μόνο ε, ε, κάτι το οποίο καταγράφει αυτά τα οποία λέγονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις. Γιατί το 2016 είχε υψηλότερη επίσημη αναπτυξική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη από ποτέ. Βλέπουμε ότι έχουμε τα κόστη των προσφύγων στις χώρες και η μεγάλη επιτυχία της Γερμανίας είναι ότι συμμετέχουν στο κλαμπ των χωρών που επίτυχαν το στόχο του 0,7. Και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι πάνω από το 1 πέμπτο της επίσημης αναπτυξιακής της βοήθειας δαπανάται πράγματι στην υποδοχή των προσφύγων. Η απονομαζόμενη λοιπόν διευκρίνηση των ε, κόστων των προσφύγων στον ΩΣΑ είναι κάτι που καλωσορίζουμε και ελπίζω να είναι τόσο συντηρητική όσο είπατε κύριε Σίτε. Θα πρέπει να είναι πολύ συντηρητική και πολύ περιοριστική. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν κάτι που με προβληματίζει εδώ καιρό. Η Επιτροπή φυσικά Ντάκα ε, του ΩΣΑ ε, έχει και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος τακτικό μέλος, ε, τακτικό μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ομάδες εργασίας όπως στατιστικών στοιχείων και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει και τη θέση της αντιπροεδρίας ε, στην τάκτη ε, του ΩΣΑ. Ποια είναι λοιπόν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες είναι οι προτάσεις της, οι θέσεις της όσον αφορά αυτή τη συνάντηση της 10ης Ιουλίου όπου θα αποφασιστεί η διευκρίνηση του, ε, του ορισμού του κόστου των προσφύγων. Ποιο θα επηρεάσει τι, τι ρόλο θα παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη συζήτηση και η Επιτροπή μας. Ε. Δεύτερον, ήθελα να πω ότι μα ανησυχεί δικαίω ε, όταν βλέπουμε ότι με αυτά τα ένα νούμερα παρατηρούμε ότι το μερίδιο για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε συρρυκνώνεται. Μα ανησυχεί ακόμη περισσότερο το γεγονό ότι η Ποσαχάρη Αφρική λαμβάνει ακόμη λιγότερα από όσα παλιότερα. Εντελώ παράλογο είναι όλο αυτό, αν σκεφτεί κανεί ε, τι ε, προκλήσει ε, για την ανάπτυξη. Η επερχόμενη είναι Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Δεν πρέπει να επαναλάβει το ποσοστό του 0,7%. Πολλέ πολιτικέ ομάδε αποφάσισαν να απόσχουν από αυτή την ψηφοφορία. Διότι δεν πρόκειται, να υπά... πρόκειται για συνένεση. Κάποιοι θα συμφωνούν, όχι όλοι. Δεν πρέπει να οδηγήσουμε την αναπτυξιακή μα συνεργασία σε μια κατάσταση όπου κάθε φορά θα λέμε ότι αντιμετωπίζουμε τι ρίζε τη μετανάστευση. Τι θα κάνει όσα με αυτή τη νέα τάση, όπου κάθε νέο εργαλείο ε, του βάζουμε πάνω μια ετικέτα, αντιμετωπίζουμε τις ρίζες της μετανάστευσης. Ευχαριστούμε κύριε Ζέλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάποιος είχε πει να εμπιστεύεσαι μονάχα τις στατιστικές που έχει παραποιήσει εσύ ο ίδιος. Τι κρύβεται άραγε πίσω από τις στατιστικές. Τεχνική απόδοση, απόδοση προσωπικού, επιδοτήσεις, δάνεια, πρόκειται για μια δέσμη δυνατοτήτων που κρύβεται ενδεχομένως πίσω από όλα αυτά τα στατιστικά νούμερα. Δύσκολο να εκφραστεί με ένα μονάχα ποσοστό. Από την άλλη μεριά δαπανώνται και σημαντικά ποσά. Μας το εξηγήσατε άλλωστε αυτό εσείς οι ομιλητές που ωραίουν σε πολλές από τις χώρες αυτές και για ορισμένες οφείλω να ρωτήσω μέχρι τώρα τι έγινε με τα λεφτά αυτά και τι μπορεί ενδεχομένως να επιτευθεί ακόμα εν ώψη των ε, πολιτικών συνθήκων σε ορισμένες από τις χώρες αυτές. Και πολύ συχνά φοβούμε ότι τα χρήματα αυτά χάνονται στις αβάνες και στις ερήμους. Αν συμπεριληφθούν τα χρήματα που έχει δώσει και η χώρα μου στην ODA, πάνω από 30 δισεκατομμύρια από δημόσιους πόρους τα τελευταία χρόνια. για την υλική στήριξη των προσφύγων. Πρόκειται για χρήματα περισσότερα από αυτά που διαθέτουν στον εθνικό τους προϋπολογισμό ορισμένες χώρες και θα πρέπει να λυθεί υπόψη αυτό. Ευχαριστώ. Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την έκθεσή σας. Δύο σύντομες παρατηρήσεις και μία ερώτηση. Αφενός, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ODA καθώς και για τη σύντομη αναφορά της Κομισιόν για τα νούμερα της ODA. Στην έκθεση δίνεται ένα πλαίσιο για το τι έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει κάνει στους διάφορους τομείς της χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Είναι καλό λοιπόν που υπάρχει αυτή η σύντομη έκθεση και που έχει δημοσιευτεί. Αλλά δεν αντικαθιστά την έκθεση για την, για την χρηματοπιστωτική ανάπτυξη που θα έπρεπε να είχαμε λάβει και την οποία δεν έχουμε πλέον. Και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να γνωρίζουμε πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών τη. Για παράδειγμα, για το χρέος των χωρών αυτών, για τη χρηματοδότηση ε, έργων για το κλίμα. Στο νέο κόνσεπτ λένε ότι θα υποβάλλονται αναφορές. Ελπίζω ότι αυτό το νέο reporting δεν θα υπολείπεται του παλαιού. Δεύτερη σύντομη παρατήρηση. Επειδή έχουμε και εκπρόσωπο της Κομισιόν και της ΔΑΚ Θέλω να σας ανακοινώσω ότι στην Επιτροπή Ανάπτυξης έχουμε αρχίσει να συζητούμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην ΤΑΚ. που έχει αναλάβει και ρόλο αντιπροεδρίας στην ΤΑΚ και έχουμε προκειμένου ορισμένες ερωτήσεις τις οποίες θα υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια τις απαντήσεις σας. Και μια ερώτηση τώρα που θα συμπληρώσω σε όλα αυτά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Αυτή η peer review για την Ευρωπαϊκή Ένωση επίκειται πάλι. Η αξιολόγηση των ομοτήμων δηλαδή. Γι' αυτό ρωτώ με ποιον τρόπο θα ζητήσετε να λάβετε εισρωές και από τη δική μας εδώ Επιτροπή Ανάπτυξης. δεύτερη σύντομη ερώτηση. Σημείωσα εκεί που είπατε προς τα που βαδίζει η ODA ότι η ελάφρυνση του χρέους δεν φαίνεται πλέον να παίζει κανένα ρόλο αντίθετα με όσα λέγονταν και συνέβαιναν στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Πού βρισκόμαστε λοιπόν, εσείς τώρα Τζούντι, τελευταία, αλλά όχι έσχατη. Ευχαριστώ για την επισκόπηση και τις διαφάνειες. Θα μπορούσαν όμως να είναι πιο ξεκάθαρα ακόμα, διότι αν κατάλαβα καλά, όλοι βλέπουμε με ικανοποίηση ότι οι δαπάνες για την ODA έχουν αυξηθεί. Βλέπουμε όμως ένα μεγάλο ποσοστό δαπανών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες DAC, για αυτούς που ζητούν άσυλο. Εμείς οι Ολλανδοί το 23% της ODA μας το δώσαμε το 15-16 για την ε, περίθαλψη προσφύγων. Άρα δαπανώνται μέσα στις ίδιες τις χώρες για ζητήματα ασύλου και σε ορισμένες Χώρε χαμηλού εισοδήματο, ιδίω αυτέ που βρίσκονται γύρω από την Συρία, εννοείται. Ενώ βλέπουμε την Αφρική και την υποσαχάρια Αφρική ιδίω, εκεί οι δαπάνε να μειώνονται. Ενώ το προσφυγικό είναι ένα σύνολο και θα πρέπει να το δούμε. Διότι μεταφέρουμε ODA από την Αφρική σε άλλε χώρε γύρω από τη Συρία, σωστό πρέπει να γίνει αυτό, μετακινούμε όμως τα ποσά αυτά από την υποσαχάρια Αφρική σε άλλες χώρες βορειότερα, που βρίσκονται βέβαια πάνω στην οδό της μετανάστευσης, να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, αλλά το είδαμε και στο, στην έκθεση του ΟΣΑ. Βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση για την υποσαχάρια Αφρική μειώνεται και η χρηματοδότηση για τις ε, χώρες της ε, Μαγκρέμπ αυξάνονται. Όλα αυτά στρέφονται γύρω από την μετανάστευση. Σωστό. Θέλω λοιπόν να πω καθαρά τα πράγματα αυτά και δυνατά. Ερώτηση τώρα. Τι ακριβώς προσπαθούμε να διευκρινίσουμε μέσα στην ΤΑΚ του ΟΟΣΑ. Όπως είπατε εσείς κύριε, είδαμε δηλαδή ότι οι κανόνες που έχουμε είναι απειρχιωμένοι και πρέπει να επικαιροποιηθούν. Τι είδους επικαιροποίηση εννοούμε. για να διατηρηθεί το επίπεδο δαπανών, για να αυξηθεί το επίπεδο δαπανών που θα προτιμούσα εγώ, τι μπορούμε να αναμένουμε. Ερώτηση όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ξεκινώντας από αυτό που, ρώτησε η κυρία Χάουταλα αλλά και η διπλανή της, ποιες είναι οι βλέψεις μας, τι, τι, πώς τα βλέπουμε δηλαδή αυτά. Τον Φεβρουάριο ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα purpose code το οποίο θα αναφέρεται ακριβώς στη μετανάστευση. Μπορείτε να μας δώσετε τους ε, κώδικες αυτούς και όχι απλώς ένα μήνυμα που να λέει ότι τον ε, διαδηλώνουμε. Διότι θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε για την εντολή που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις της ΔΑΚ. Δεν την ε, βλέπουμε την εντολή αυτή και αυτό με ενισχύει πολύ. Και ερώτηση προς τον εκπρόσωπο του ΟΣΑ. Μπορείτε να διευκρινίσετε περισσότερο ποιοι είναι οι στόχοι σας με αυτή την επανεξέταση των ε, ε, δαπανών για την ΤΑΚ. Θα συζητήσουμε τη στρατηγική για την Αφρική και τη νέα εταιρική σχέση που είναι ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε την μετακίνηση της βοήθειας και τη βάζουμε επιτάπητος και θα χρειαστούμε να έχουμε και feedback από την συνάντηση των Υπουργών που έγινε στις 19 Μαΐου. Να λοιπόν, ήταν ξεκάθαρες οι ερωτήσεις. Ας αρχίσουμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία μου. Ίσως με τα θέματα που ρώτησαν πολλοί για την διαφάνεια της εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν πηγαίνει στον ΩΣΑ. Τι περιλαμβάνει η εντολή αυτή. Ή μήπως προτιμάτε να αλλάξουμε πάλι τη σειρά, δηλαδή να μιλήσει ο κ. Σιούτε. Α, κυρία Μέρλο πρώτη λοιπόν, σύμφωνη. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με την αξιολόγηση της εργασίας που γίνεται ε, με τις ε, δαπάνες προσφύγων στις δωρήτριες χώρες που έχουμε εδώ έχει γίνει εργασία βεβαίως από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας και βλέπουμε τι είναι επιλέξιμο, τι δεν είναι επιλέξιμο και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει διαφήνεια, διαφάνεια, συγκρισιμότητα. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε καλύτερα πώς θα γίνει αυτή η εργασία, διότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, σαφείς ε, τι μπορεί να είναι επιλέξιμο για επίσημη αναπτυξική βοήθεια και θα πρέπει να αυξήσουμε την συγκρισιμότητα και την διαφάνεια των δαπάνων, δαπανών που καλύπτονται. θα πρέπει να υποστηρίξουμε βεβαίως και τις ίδιες τις χώρες. Αυτό είναι κάτι τα πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή και εμείς θέλουμε συμμετοχή με τις χώρες μέλη ε, για να αυξήσουμε τη συμμετοχή στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να έχουμε και προβλέψεις. Είναι πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε σε σχέση με το στόχο, αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι χώρες αυτές τι μπορούν ε, να ε, έχουν, να προβλέψουν, ε, να έχουν προσδοκίες για το τι θα έχουν. Τα κράτη-μέλη βεβαίως είναι υπεύθυνα για τις δεσμεύσεις αυτές και αυτό εξαρτάται από τις δημοσιονομικές τους αποφάσεις. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό. Ε, ίσως αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τις χώρες. Υπάρχει υποχρέωση από τις συνθήκες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αποτελέσματα, να ε, συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη, να προγραμματίζει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ίσως πρέπει να γίνει εργασία, ίσως όχι στη δική σας υπηρεσία της Επιτροπής, αλλά σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλα τμήματα. Ίσως ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να αναφέρω έχει, έχει σχέση με την λογοδοσία, την έκθεση λογοδοσίας. Η παρακολούθηση είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη για να βεβαιωθούμε ότι έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις και η όλη διαδικασία στο πλαίσιο αυτό αξιολογούμε το σύστημα ε, υποβολής εκθέσεων ούτως ώστε να ε, δούμε αν αυτό είναι συμβατό με την ατζέντα της Αντίσα και το πρόγραμμα 2030. Όπως ξέρετε, ε, φέτος δεν είχαμε τέτοια έκθεση. Τώρα έχουμε όλα τα στοιχεία ε, το περιεχόμενο του πλαισίου αυτού για την ατζέντα και μεταφράζουμε ε, στην υπηρεσία μας ε, το, την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κοινοποίηση αυτή και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε, να μην υπάρχει επικάλυψη με άλλες εκθέσεις. Βεβαίως θα επαναλάβουμε αυτή την έκθεση, είναι δέσμευσή μας και βεβαίως θα έχουμε το ίδιο πεδίο εφαρμογής, το ίδιο εύρος. Ε, θα, θα έχουμε παρόμοια κάλυψη, αλλά μέσα σε νέο πλαίσιο. Ναι, στο τέλος να μιλήσετε. Βλέπω ότι αυτοί που έθεσαν ερωτήσεις ε, πρέπει να πάω στην Επιτροπή την ε, νομική Γι' αυτό δεν άκουσα να απαντήσατε τις ερωτήσεις για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με την διευκρίνηση αυτών των Indonor Refugee Costs. Ξέρετε ότι η Επιτροπή έχει έναν κώδικα DAC ε, στην Επιτροπή Στατιστικής στις 28 ε, Φεβρουαρίου. Θέλουμε τη θέση αυτή που είπα ότι θα διευκρινίσει η Επιτροπή. Ίσως στο τέλος, εσείς στο τέλος. Να, ε, επειδή η κυρία πρέπει να φύγει, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πιστεύω θα μιλήσει γι' αυτό και ο συναδελφός μου. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Σκοπός αυτού του εργαλείου. Συγγνώμη, δεν σας ρωτούν για τις λεπτομέρειες. Όσα δουλεύει για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που σας ρωτάνε, αυτό που σας ρωτάει η συνάδελφος είναι ποια θα είναι η απόκριση της Κομισιόν. Προετοιμάζετε, πώς προετοιμάζετε την ε, εργασία σας γι' αυτό. Δεν ακούγεται δυστυχώ η ομιλήτρια. Δεν ρωτάμε τι δουλειά κάνει ο ΩΣΑ, αλλά πώς προετοιμάζει τη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διαπραγματεύσεις. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Οπότε κυρία Μερλό, ε, τι γίνεται, επειδή είναι ε, στο δικό τους πεδίο αρμοδιότητα, αν όχι πρέπει να βρούμε σε ποιον; Ε, όχι απόλυτα, απαντάει κυρία Μερλό. Ωραία λοιπόν, θα το συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε να το διερευνούμε, θα ψάξουμε να βρούμε πώς λειτουργεί, οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Σούτερ Για τη μετανάστευση. Να πω ότι πρόκειται για μια σύνηθη πρακτική για μας. Διάφορα μέλη προτείνουν ε, κώδικες ε, που εγκρίνονται μετά από τη γραμματεία και τα μέλη για τη μετανάστευση παρουσιάστηκε στην άτυπη συνάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο και θα ξαναπαρουσιαστεί σε μια επίσημη συνάντηση μέσα Ιουνίου. Τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου θα επισημοποιηθεί η υποβολή της πρότασης αυτής. Αν ξέρω τι ακριβώς κάνει η Κομισιόν, όχι. Υπάρχει διαδικασία και συνεχίζεται. Τώρα για το ερώτημα του κύριου Λίτς, ε, γιατί αποτελεί κομμάτι της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, υπάρχει εδώ και 35 χρόνια σχεδόν, από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Ε, τώρα γίνονται συζητήσεις για τη λογική στην οποία βασίζεται. Υπάρχουν διάφορε λόγοι, ανθρωπιστική, αναπτυξιακή, ασφάλεια, παγκόσμια. Και τώρα είναι σαφές ε, ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση με την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική πτυχή στο πλαίσιο της πενταετίας αυτής. Ε, θα αποτελεί λοιπόν και θα συνεχίσει να αποτελεί κομμάτι της ε, επίσημης ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά θα καθοριστεί, θα ορίζεται πιο συγκεκριμένα από ότι τα τελευταία χρόνια. Εμείς θεωρούμε ότι και τα νούμερα που θα υπάρξουν θα το θα τεκμηριώσουν αυτή την προσέγγιση. Τώρα είπατε τι είδου κανόνες. Ε, εγώ ασχολούμαι με τους κανόνες υπολογισμού. Ε, ε συγγνώμη, του κανόνε που ορίζουν ότι κάτι εντάσσεται στην επίσημη αναπτυξική βοήθεια. Μετά πρέπει να δούμε ποιε θα, ε, θα είναι οι συνέπειε ε, όσον αφορά τη μεταναστευτική κρίση και πώ μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα εργαλεία. Αυτή θα είναι η δεύτερη φάση του έργου μα. Κάτι που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η ομάδα εργασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι τέλη του έτου. Αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί στο πλαίσιο ενό άλλου θέματο ενδεχομένω, ε, αλλά δεν πρέπει να το ρωτήσετε για μένα, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα δική μου. Αλλά είναι κομμάτι των εργασιών που γίνονται αυτή τη στιγμή. Κάποιο είπε ότι το σύστημα έχει αποτύχει το παρελθόν, κοιτάτε λέγοντα αυτό. Ε, αυτό δεν μα βοηθά να κοιτάμε το μέλλον. Ναι. Προφανώ υπάρχει η διαφάνεια, η λογοδοσία τα λαμβάνουμε υπόψη στις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Θα γίνει και μια έρευνα δαπανών ώστε να έχουμε μια αίσθηση του πού θα πάνε τα πράγματα μέσα στην επόμενη διετία, τριετία. Για να απαντήσω την ερώτησή σας για την ευρύτερη εικόνα του τι θα έχουμε επιτύχει το 2020, αν θα έχουμε επιτύχει το 0,7%, δεν το γνωρίζω. Πάντως, συναδέλφοι, που πραγματοποιούν αξιολογήσεις μεταξύ ομοτήμων ε, παρατηρούν ότι τα κράτη-μέλη έχουν σαφείς στρατηγικές για να αυξήσουν το ποσοστό τους μακροχρόνια μέχρι το 2030 όσον αφορά την αύξηση του, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν αναφέρεται ακριβώς που θα γίνει, αλλά θα γίνεται, αξιολόγηση, γίνεται αξιολόγηση σε βάθος. Ε. says, well, is, is this, uh, Mr. Ο κύριος Ζέλα ε, ε, αναφέρθηκε σε ένα θέμα που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, και την υποσοχαρή Αφρική. Είναι θέμα διαφάνειας και όλες συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Είναι Δύσκολα θέματα για όλους μας. Αυτό που μπορώ εγώ να σας δώσω είναι πια μια, απλώς μια λεπτομερή εικόνα του ποιος ξοδεύει ανατομέα σε κάθε χώρα υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία και αυτό βοηθά και τις χώρες ε, δικαιούχους ε, να αποδώσουν ευθύνε. Ε, μπορούν να μας πούνε, μας υποσχεθήκατε τόσα χρήματα, πού πάνε αυτά τα χρήματα και μετά οι προσπαθίες μας επίσης εστιάζονται στη βελτίωση όλων αυτών. Μετά μιλήσαμε για την ελάφρυνση του χρέου που προέκυψε το 2016. Διαρκώς παρατηρούμε αυξομοιώσεις αλλαγές μάλλον στο, όσον αφορά την ελάφρυνση των χρεών. Είχαμε το 2016 την Κούβα, την Ισπανία, λόγω του γεγονότος ότι η Ισπανία παρήχε σημαντική ελάφρυνση χρέους προς την Κούβα. Έγινε μια ερώτηση για την ε, ε, αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων και τι σχέδια έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ε, συνάδελφο ασχολείται με αυτό, οπότε θα το στείλω εκεί. Αυτά όσον αφορά τι ερωτήσει ε, που μου απευθύνει το κοινό. Ε, θα δούμε το πώς η Κομισιόν προετοιμάζει το θέμα κάποια άλλη στιγμή. Για το, θα βρούμε τον αρμόδιο εκεί. σε κάποια μελλοντική συνάντηση. Σάρλ, θέλετε κάτι να πείτε πριν κλείσουμε. Όχι δεν, θέλω, δεν έχω τίποτα εναντίον του ομιλητή της ομιλήτριας για να είμαι σαφής. Αυτό το οποίο κατηγορώ εδώ είναι η έλλειψη μεθόδου. Έχουμε 0,7% που αφιερώνεται στο σκοπό αυτό και εδώ και τόσα χρόνια δεν λειτουργεί το σύστημα. Εγώ αυτό το οποίο ζητώ είναι η Κομισιό να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, να στριμώξει τα κράτη-μέλη και να τα καλέσει να κοινοποιήσουν ε, τα στοιχεία το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι εφικτό διότι μπορεί κανείς αυτό να το δει στις, στους προϋπολογισμούς που δημοσιεύονται στις επίσημες εφημερίδες των κυβερνήσεων. Αυτό που λείπει είναι η προβλεψιμότητα, η προοπτική. Τα κράτη-μέλη μιλούν για τα πάντα, και δεν μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να τηρήσουν τις ε, δεσμεύσεις τους. Είναι κοροϊδία αυτό. Είναι εδώ χρόνια και χρόνια που προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τα πράγματα, δεν έχουμε καμία αντίδραση και είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα ψηφίσω το κονσένσου στο ευρωπαϊκό για την ανάπτυξη. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κοροϊδία, αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει τα κρατημέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μας πούν σαφώς, όπως κοινοποιούν τα στοιχεία τους στην Κομισιό, τα στοιχεία τους στα δημοσιονομικά τον Οκτώβριο κοινοποιούν το σχέδιο προϋπολογισμού ε, για το επόμενο έτος, δηλαδή τον Οκτώβριο 2007, θα λάβει η Κομισιόν τα σχέδια των προϋπολογισμών, τα οποία περιλαμβάνουν την αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης, τα κράτη-μέλη κοινοποιούν ε, τις εκτιμήσεις για τα τρεις, τους τρεις επόμενους προϋπολογισμούς. Εφόσον ξέρουν την προβλέψεις ε, για τις τρεις επόμενες χρήσεις επειδή αντιστοιχούν ε, στην ε, υποχρέωση να είναι πιο σαφής, γιατί να μην μας κοινοποιούν επίσης αυτό που προβλέπουν στις εκτιμήσεις της δημοσιονομικές για τις τρεις επόμενες χρήσεις. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν για να μην έχουμε καμία αμφιβολία για το τι θα πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σταματήσουμε αυτό το συλλογικό ψέμα που είναι απαράδεκτο. Περιμένω λοιπόν η Κομισιό να, να διαβιβάσει την επιθυμία αυτής της υπηρεσίας στον Επίτροπό σας και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, διότι περνάνε χρόνια και χρόνια και θα φτάσουμε στο 2030 και θα ανανεωθεί η δέσμευση που απέτυχε το 2005 και το 2015. Ναι. Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά όλες αυτές τις εξελίξεις και πώς εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον ΩΣΑ, ποιες θέσεις υποστηρίζει. Θα γράψουμε και στον Επίτροπο να ρωτήσουμε για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ και εσάς κυρία Μέρλο και εσάς κύριε Σούτε και είναι βεβαίως τα θέματα αυτά κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Okay, colleagues, we have, we're running behind time now, and I do want to... Κάπως έχουμε καθυστερήσει. Πρέπει να προχωρήσουμε γιατί μας περιμένει και η ψηφοφορία. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο. Έχουμε όμως ένα σημαντικό θέμα, το, το 7, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και στην ειρήνη με γνωμοδότηση για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Τη συντάσσουμε εμεί δηλαδή για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, για την τροποποίηση του κανονισμού για το μηχανισμό συμβολή στην σταθερότητα και στην ειρήνη. Το θέμα αυτό βέβαια δεν είναι και ε, ε, δεν βρίσκει μάλλον όλους απολύτως σύμφωνους, γιατί υπάρχουν 75 τροπολογίες. Χωρίς όμως να μακρηγορήσω περισσότερο, θα δώσω το λόγο στον Πάβο Βάιρινεν, που είναι ο εισηγητής της γνωμοδότησής μας και θα μας εξηγήσει πού βρισκόμαστε και πού οδηγούν τα επόμενα βήματα. Κυρία Πρόεδρε, βεβαίως η πρόταση σε ένα βαθμό είναι αμφιλεγόμενη, όπως εξήγησατε. Από την άποψη όμως της Επιτροπής Ανάπτυξης φαίνεται να επιλέγουμε μια κοινή προσέγγιση για το σχέδιο αυτό κανονισμού. Για μας, βέβαια, είναι σημαντικό το ερώτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί χρηματοδότηση για το μηχανισμό αυτό και μας ενδιαφέρει και η χνηλασιμότητα της ε, χρηματοδότησης. Στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως που έχω συντάξει προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα και να αντιμετωπίσω τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί, προβλέποντας και μια προσθήκη που λέει ότι δράσεις για capacity building θα εγκρίνονται στην βάση των κριτηρίων της ODA που θεσπίζει ο OSA, DAC, DAC δηλαδή. Capacity building, δημιουργία δυναμικού, σημαίνει των στρατιωτικών δυνάμεων των ε, χωρών εταίρων. Τονίζω ότι η διατύπωση αυτή περιορίζει τον όρο αυτών στο capacity building, στη δημιουργία δυναμικού. Δηλαδή, για άλλους σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, χρηματοδότηση που να μην είναι DACable, που να μην υπάγεται στην DAC δηλαδή. Όμως, για τη ε, δημιουργία δυναμικού, capacity building, πρέπει να υπακούει στους κανόνες αυτούς. Υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα που έχει προτείνει η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Να αποκλείσουμε δηλαδή την χρηματοδότηση DCI του μηχανισμού. Αυτές είναι οι δύο δυνατότητες. Εγώ προτιμώ την δική μου πρόταση για τους εξής δύο λόγους. Πρώτο, θεωρώ ότι ο συνδυασμός και πα και αναπτυξιακής χρηματοδότησης είναι μια καλή λύση, γιατί δίνει μια θετική, υπαγορεύει μια θετική πορεία. Δεύτερο, μπορούμε να διαθέτουμε περισσότερους πόρους υπέρ του μηχανισμού εάν χρησιμοποιηθεί και χρηματοδότηση DCI. Μπορώ να δεχτώ όμω και την πρόταση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Απλώ εκδηλώνω την προτίμησή μου υπέρ τη δική μου. Διεξήχθη συνάντηση των σκιωδών τη Επιτροπή Εξωτερικών. Ανησυχούσα για εκείνη την συνάντηση, διότι γνωρίζαμε ότι ο συνάδελφός μας Ντανζάν είχε συντάξει σχέδιο έκθεσης για λογαριασμό της ΑΦΕΤ οι τροπολογίες της οποίας, για την οποία έκθεση δηλαδή, θα καθιστούσαν το αποτέλεσμα μη αποδεκτό από πολλές απόψεις για μας. Στη συνάντηση αυτή, ο Τανζάν παρετήθηκε από τη βασική του πρόταση δεν ζητεί πλέον αντικατάσταση των έκτακτων ή exceptional circumstances περιστάσεων από ειδικέ special, ούτε προτείνει αλλαγή των υποπαραγράφων α και β η λέξη και να αντικατασταθεί από τον διαζευτικό σύνδεσμο ή. Άρα παρετείται από τις βασικές του προτάσεις. Συζητήσαμε ακόμα και τις δύο εναλλακτικές επιλογές πώς να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες της Επιτροπής ΔΕΔΕ και είπε ότι η πρόταση σοσιαλιστών και δημοκρατών μπορεί να εξεταστεί. Είπε επίσης ότι και η δική μου πρόταση μπορεί να εξεταστεί. Δεν ξέρω σε ποιο συμπέρασμα έχει καταλήξει. Πάντως φάνηκε εύκαμπτος και επικοδομητικός. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση που να είναι ικανοποιητική και για μας. Αύριο θα διεξαχθεί νέα συνάντηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών της ΔΕΒΕ και τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες, καθώς και τις δύο αυτές εναλλακτικέ επιλογές που σας εξήγησα. Ευχαριστώ. Άρα δηλαδή σημειώθηκε κάποια πρόοδο στις θέσεις των δύο επιτροπών από την τελευταία μα συνεδρίαση και εντεύθεν. Ο κύριος Βέντε. Ε, εκ μέρους του κύριου Κόγκα και όδους του ΕΛΚ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Υποστηρίζουμε απόλυτα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι υπάρχει ανάγκη συγκεκριμένης δράσης για την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων ε, στις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως έχω τονίσει ήδη στην Επιτροπή μας, ε, η ασφάλεια ε, είναι βασικό ζήτημα. Πρέπει να συντονίσουμε τις δράσεις μας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα της ανάπτυξης ε, και για να επιτύχουμε τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Η θέση της ομάδας μας είναι σαφής. Θέλουμε το εργαλείο αυτό, το μηχανισμό αυτό, θέλουμε να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό. Δεν θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε περαιτέρω αιρεσιμότητα. Επίσης πιστεύουμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να ζητάμε ε, να έχει τις πλήρες δυνατότητες δηλαδή, μηχανισμό, ο μηχανισμός αυτός διότι αυτό θα υπονομεύσει την ελαστικότητά του. Ωστόσο, υποστηρίζουμε την ιδέα ότι η χρηματοδότηση που υπάρχει ήδη δεν πρέπει να αναπτυχθεί, να μην δοθούν δηλαδή αυτά τα χρήματα σε αυτό το μηχανισμό. Αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σιγητή για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει για να συνομιλήσουν οι ομάδες μας ε, για το θέμα αυτό, αλλά και για να συνομιλήσει στην Επιτροπή Άφετη για το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό που δείχνει ελαστικότητα όσον αφορά τις τροπολογίες. Και εγώ εδώ χαίρομαι ιδιαίτερα που το ΕΛΚ υποστηρίζει τη δική μου πρωτοβουλία. Η DCI δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό το μηχανισμό θα άλλαζε κατεύθυνση. Οπότε αν βγει η DCI μπορούμε να έχουμε αυτό το μηχανισμό και έχω υποβάλει σχετικέ τροπολογίες, Θα πρέπει να έχουμε ένα θετικό κατάλογο ιδεών. Τι μπορούμε να υποστηρίξουμε ως μηχανισμό. Και εμείς πιστεύω ως κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Δεν ε, δεν, έχει, δεν έχουμε αναλάβει δρασει για τα καταπιστεύματα για την Αφρική, δεν έχουν γίνει ενεργά βήματα, οπότε το κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να πει σαφώς τι υποστηρίζει και να δώσει τα εργαλεία στην Κομισιόν. Εξακολουθώ λοιπόν να είμαι υπέρ και προσβλέπω στις συζητήσεις μας ε, να δούμε κατά πόσο η DCI μπορεί να βγει από αυτόν τον προπολογισμό Πολλές ΜΚΟ ε, σε όλη την Ευρώπη έρχονται σε επαφή μαζί μου για αυτό το θέμα και αυτό είναι σαφές μήνυμα από την κοινωνία των πολιτών. Να μην αναμειγνύουμε τα θέματα. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Χόκερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Επειδή δεν είναι παρούσα συναδελφός μου, θα μιλήσω εξ ονόματος των Πρασίνων. Να ευχαριστήσω πρώτα τον Πάγο Βάιρινεν για την ε, γνωμοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω άνοιξε την πηξίδα της Πανδώρας. Μας υποβάλλει μια πρόταση για τον μηχανισμό σταθερότητας που μέχρι τώρα προοριζόταν μονάχα για ε, μη στρατιωτικούς σκοπούς και προτείνει την επέκτασή του για την δημιουργία στρατιωτικού δυναμικού σε τρίτες χώρες με βάση το άρθρο 209, το οποίο προβλέπει ωστόσο πολιτική ανάπτυξη. Έχουμε φτάσει λοιπόν τώρα σε ένα σημείο όπου πολλέ χώρε μέλη και η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας οδηγούσαν εδώ και καιρό. Δηλαδή, έχουμε για τόσο πολύ καιρό δηλώσει και επικοινωνήσει και δεχτεί τέτοια διαρκή πειρά για την σύνδεση αυτή μεταξύ των πολιτικών, ώστε επιτέλους να εγκρίνουμε στρατιωτικές δαπάνες και να χρηματοδοτούνται αυτές μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για ένα, ε, ε, ένα μόρφωμα το οποίο στέκεται ωστόσο πάνω σε πολύ ασταθή πόδια και οι τρεις νομικές υπηρεσίες και του Συμβουλίου και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου λένε ότι έχουν σημαντικότατες αμφιβολίες σχετικά με την νομιμότητα της πρότασης αυτής. Τώρα, έχω να σας πω τα τρία εξή. Το άρθρο 41 της συνθήκης απαγορεύει χρηματοδότηση επιχειρήσεων στον στρατιωτικό τομέα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αποτελεί την συμβατική μας βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο 40 δε, λέει καθαρά ότι η εκτέλεση της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας δεν γίνεται σε βάρος άλλων πολιτικών. Και αυτό είναι λοιπόν μια πολύ ξεκάθαρη δήλωση. Υπάρχει και καθαρή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι προτάσεις οι οποίες έχουν τη βάση τους σε ένα άρθρο της συνθήκης οφείλουν να οδηγούν σε εφαρμογή της προβλεπόμενης, στο άρθρο αυτό, πολιτικής γιατί αλλιώ θα μπορούσαμε να πάρουμε χρήματα από την αγροτική πολιτική για να χρηματοδοτούμε δράσει κατά τη τρομοκρατία. Στην προκείμενη περίπτωση πρόκειται για ένα αγαθό το οποίο προβλέπει την πολιτική ανάπτυξη και επομένω πρέπει να συζητεί ζητήματα ανάπτυξη και όχι στρατιωτική ασφάλεια. Βλέπω ξανά και ξανά τα χρήματα της αναπτυξιακής πολιτικής να διοχετεύονται σε άλλες πολιτικές. Και πολύ ελαφρά την καρδία τα χειρίζεται αυτά τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και ορισμένε χώρε μέλη. Θέλω ωστόσο να τονίσω το εξή ακόμη. Εμά δεν μα ενδιαφέρει το ζήτημα τη ασφάλεια. Ε, μάλλον δεν θεωρούμε ότι το ζήτημα τη ασφάλεια δεν είναι σημαντικό. απλώ δεν θέλουμε την διασύνδεση μεταξύ πολιτική ασφάλεια και αναπτυξιακή πολιτική. Αυτή η διασύνδεση υπάρχει, αλλά η χρηματοδότηση δεν πρέπει να ανακατεύεται. Άλλοι πρέπει να είναι οι μηχανισμοί για την ε, ανάπτυξη, η χρηματοδότηση ανάπτυξη δηλαδή, και άλλοι μηχανισμοί για τη στρατιωτική ασφάλεια. Αυτό μας ενδιαφέρει εν τέλει. Δεν πρέπει να ανακατεύονται τα πράγματα στη χρηματοδότηση. Χρειάζεται ξεκάθαρος διαχωρισμός. Και βλέπουμε τελικά ότι η βιομηχανία των εξοπλισμών ασκεί επιρροή διαρκώς εδώ. Θέλω δεν επισημάνω ακόμη ότι η πολιτική ασφάλειας, την οποία ως πράσινη την δεχόμαστε, ξαναλέω, δεν μπορεί ωστόσο να αποβεί σε βάρος της χρηματοδότησης των σχολείων, της παιδείας, της περίθαλψης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ποιον υποστηρίζουμε στην περίπτωση αυτή στην Αφρική, θα πρέπει να είναι σαφές ότι και τα όργανα ασφαλείας εκεί δεν διαθέτουν την παράδοση να εμφανίζονται και να είναι, δηλαδή να παίζουν το ρόλο των προστατών των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Όπως τα κατανοούμε τα πράγματα αυτά εμείς. Εν τέλει, χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση των μηχανισμών ασφαλείας στις χώρες αυτές χρειαζόμαστε επαρκή κοινοβουλευτικό έλεγχο και από τη δική μας πλευρά αλλά και από τα κοινοβούλια των ενδιαφερομένων χωρών. Και το βρίσκω λυπηρό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά και ξανά τα παραμιλεί τα πράγματα αυτά. Υποστηρίζουμε τη γραμμή του εισηγητού εν τέλει. Οι πόροι θα πρέπει να σέβονται τις κατευθύνες γραμμές του οοσα θα πρέπει λοιπόν να είναι πολύ ξεκάθαρη γραμμή και τη γραμμή αυτή την έχει ήδη δείξει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, τέρες Ναι, ευχαριστώ. Ίσως να μην κατάλαβα καλά κάτι. Εγώ να πω ότι είναι συμφωνώ με το ότι πρέπει να γνωρίζει κανείς την ακριβή προέλευση των κονδυλίων. Ωστόσο, για τους στόχους της ε, ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ήμουν στα Ηνωμένα έθνη και ακούγα διαρκώς να αναφέρεται αυτός ο στόχος ειρήνης και ασφάλειας και ισχυρών θεσμών. Διαρκώς ε, γινόταν αναφορά στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη και πριν δύο χρόνια έγινε μια ακρόαση εδώ για την ανάπτυξη και την ασφάλεια και σίγουρα αιτιολογείται. Το, το συζητάμε. Κονδύλια λέμε για την ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι λογικό. Ωστόσο, δεν πρέπει να αφαιρέσουμε χρήματα από την καταπολέμηση της φτώχειας ή την υποστήριξη της εκπαίδευσης για να τα δώσουμε στην ασφάλεια σε καμία περίπτωση. Οπότε εσείς μιλάτε για την έννοια της ασφάλειας που έχουμε και ότι οι έννοιες ασφάλειας για μας είναι διαφορετικές ε, από τις άλλες χώρες. Για μένα ασφάλεια σημαίνει πολύ απλά ότι τα κορίτσια για παράδειγμα μπορούν να πάνε στο σχολείο χωρίς να τα απαγάγει κανείς ή να τα βιάσει κάποιος ε, και μετά από δύο χρόνια να μην ξέρει κανείς που βρίσκονται ή όπως στην Αίγυπτο να επιτίθεται κάποιος σε ένα πούλμαν σε κοριτσάκια που πηγαίνουν για προσκύνημα. Ε, αυτό είναι θέμα ασφάλειας και μετά παραπονιόμαστε και λέμε δεν ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα γιατί δεν υπάρχουν ισχυροί θεσμοί, δεν ξέρουμε τι έγιναν με αυτά τα χρήματα, ε, αν χρηματοδοτήθηκε η τρομοκρατία. Ε, ή ξαφνικά και μετά πρέπει να ξέρουμε περισσότερα λεφτά για τα όπλα. Είναι σίγουρα πρέπει να δώσουμε λεφτά για την ασφάλεια, αλλά ασφάλεια ε, φυσικά σημαίνει ανθρώπινη ζωή. Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Ε, ε, πρέπει να, δεν είναι δυνατότητα να πάει κανείς στο σχολείο να πεθάνει αλλά δεν πρέπει να βγάλουμε χρήματα υπέρ της ασφάλειας από, άλλα, από άλλους τομείς. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ταμείο ασφάλεια ε, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάπτυξη, ε, σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Όλοι θέλουν περισσότερη ασφάλεια, όλοι θέλουν περισσότερη ανάπτυξη και ανάμεσα στη πτώχεια και στην ανασφάλεια υπάρχει κάποια σχέση. Όταν η Γαλλία πήγε στο Μαλί, όταν οι τζιχαντιστές βρισκόντουσαν σε απόσταση 50 χιλιόμετρων από τη Μαμάκο. Ευτυχώς η Γαλλία έσωσε την τιμή της Ευρώπης, αλλά είναι ε, μια επιχείρηση που πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το προϋπολογισμό ανάπτυξης. Όλες οι χώρες που ενέκριναν την επιχείρηση στη Γαλλική θα έπρεπε να είναι συνυπεύθυνα στη χρηματοδότηση. Η Συνδίκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι υπάρχει μια διάκριση που πρέπει να γίνει. Στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής ανάμεσα συνεργασία για την ανάπτυξη και τις άλλες συνεργασίες, είτε είναι οικονομικές, εμπορικές, στρατιωτικές. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής διάκριση και νομίζω ότι αυτή η διάκριση θα πρέπει να αντανακλάται επίσης και στη δημοσιονομική πρακτική. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση. Ο κύριος Λίκ που είναι εδώ, την Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα τελείωσε η νομική επιτροπή, οπότε ε, υπάρχει προσέλευση. Ναι, ναι, ναι. Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία, λίγη ησυχία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία για την, ε, την, την σύνδεση ανάμεσα ε, στην ανάπτυξη και την ασφάλεια προς τις δύο κατευθύνσεις, διότι η φτώχεια οδηγεί στην βία, στις συγκρούσεις. Η έλλειψη ασφάλειας παρεμποδίζει ε, τις δραστηριότητες των πολιτών. Αυτό, αυτή είναι η φιλοσοφία ε, πίσω από αυτή την πρόταση. Θα πρέπει να, είναι καλό να συμφωνούμε για τις ιδέες, αλλά η πρόκληση είναι να έχουμε κάτι συγκεκριμένο επιτάπητος. Στόχος μας δεν είναι ε, να έχουμε κάτι ε, το οποίο ε, να είναι ε, το CFSP είναι για τα κράτη-μέλη μας με τα λεφτά τους και με τα χρήματά τους. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν και πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση των τοπικών ε, δυνάμεων, ούτω ώστε να, όχι για στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά για την προστασία ή αποκατάσταση του κράτους δικαίου, των κανόνων, ε, την προστασία των ε, πολιτών, των αμάχων που βρίσκονται σε ακραίες περιπτώσεις. Σε πλαίσιο τροτότητας, όταν υπάρχει βεβαίως η αστυνομία οι διοκτικές αρχές, οι ακτοφυλακές δεν μπορούν να δράσουν και πρέπει να ληφθούν μέτρα και σε πάρα πολλές χώρες σε περίπτωση κρίσης ή πρόκτη κρίση υπάρχουν καταστάσεις πολύ ευαίσθητες και θα πρέπει, χρειάζεται ενίσχυση των διοκτικών αρχών, της αστυνομίας για να προληφθεί το χειρότερο. Και αν συμβεί το χειρότερο, τότε καλούνται οι στρατιωτικοί για να αποκαταστήσουν αυτό που μπορεί να αποκατασταθεί, για να προστατεύσουν τις φυσικές συνθήκες ανάπτυξης ή να αποκαταστήσουν μια κατάσταση όπου οι αναπτυξιακοί πρωταγωνιστές, η κοινωνία των πολιτών θα βρεθούν σε κανονική, σε ομαλή κατάσταση. Βεβαίως η ΚΠΑ δεν μπορεί να κάνει τα πάντα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλές χώρες, οι στρατιώτες ε, είναι μέλος είτε μέρος της ανάπτυξης ή της διαδικασίας αποκατάστασης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Βεβαίως δεν πρόκειται να στερήσουμε την ανάπτυξη από ορισμένα κονδύλια, αλλά να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα αναπτυξιακά κονδύλια για να εκπαιδεύσουμε ορισμένες ένοπλες δυνάμεις ούτως ώστε να εκπαιδευτούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την, τα θέματα των πολιτών, για τον εξοπλισμό, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ορισμένες δράσεις στήριξης των ε, ομάδων ε, των δυνάμεων ασφαλείας. Αλλά ορισμένες φορές δεν μπορούμε να συμπράξουμε με τους στρατιωτικούς. Βεβαίως ε, έτσι δεν καταχρώμεθα τα χρήματα για αναπτύξη, της αναπτυξιακής βοήθειας για στρατιωτικούς σκοπούς. Απλώς εκπαιδεύουμε έναν άλλον πρωταγωνιστή που σε κρίσιμες καταστάσεις μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης. Και τρίτον, για ε, την ε, μείωση των ε, χρημάτων από την αναπτυξιακή συνεργασία, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για σχετικότητα. Έχουμε ακόμα για τις προοπτικές, τις δημοσιονομικές, ακόμα τρία χρόνια. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε κάτι. Για να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια από το μέσο ε, γειτονίας, από την ΚΕΠΑ, από την αναπτυξιακή συνεργασία ε, για να εκπαιδεύσουμε αυτές τις δυνάμεις ε, για να μάθουν πράττοντας, κάνοντας, πρακτικά. Στις συζητήσεις για τις μελλοντικές εξωτερικές σχέσεις θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Ε, απαντώντας ορισμένες από τις παρεξηγήσεις που άκουσα, ήθελα να κάνω αυτές τις διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε κύριο Βάρεν. Να ξέρω θα έχουμε την ψηφοφορία σε λίγα λεπτά συνάδελφα, αλλά παρακαλώ κάντε λίγο ισχύα για να ακούσουμε τον κύριο εισηγητή τον κύριο Βέρενα. Ε, ναι, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και αύριο μεταξύ σκιωδών εισηγητών. Ελπίζω λοιπόν θα καταφέρουμε να βρούμε μια καλή λύση. Δεν έχουμε ακόμα συμβαστικές τροπολογίες. Ε, ελπίζω να έχουμε αύριο. Σε κάθε περίπτωση θα συναντηθούμε και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και τις πιθανές συμβαστικές. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ να επενθυμίσω συνάδελφοι ότι θα ψηφίσουμε στις 26 Ιουνίου στην Επιτροπή μας για αυτή την νομοθετική γνωμοδότηση και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα λάβει χώρα 11 Ιουλίου και στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ωραία λοιπόν, πάμε τώρα στην ψηφοφορία. Στη μία ψηφοφορία που έχουμε. Συνάδελφοι, ξέρετε ότι αρχικά είχαμε προβλέψει να ψηφίσουμε για την Ευρωπαϊκή Συνέντευξη για την Αναπτύξη στο Στρασβούργο, αλλά δεν να ολοκληρωθεί η διαβουλεύση του Συμβουλίου, ώστε ως αποτέλεσμα δεν είχαμε τελικό κείμενο. Ε, έχουμε τώρα κείμενο που υιοθετήθηκε 19 Μαΐου από το Συμβούλιο και πλέον έχουμε ένα τελικό κείμενο το οποίο θέτουμε σε ψηφοφορία. Δεν θα ψηφίσουμε για το ίδιο το κείμενο, αλλά για ένα ψήφισμα αυτό θα συνοδεύει το κείμενο. Πρέπει να έχετε λάβει τον καταλογό ψηφοφοριών μπροστά σας. Έχουμε δύο εισηγητές, τον κύριο Νόρμπερτ Νόιζερ και τον κύριο Βέντα. Ο Νόρμπερτ Νόιζερ δυστυχώ δεν είναι μαζί μας σήμερα εδώ είχε κάποια θεραπεία που δεν μπορούσε, ιατρική που δεν μπορούσε να αναβάλει. Ο κύριος Βέντα είναι εδώ. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Βέντα πριν να ψηφίσουμε. Thank you, Linda. Ευχαριστώ Λίντα. Φυσικά θα ήθελα να πω μερικά λόγια πριν ξεκινήσουμε. Ο συναδελφός μου ο Νόρμπερτ δεν μπορούσε να είναι μαζί μας εδώ σήμερα αλλά και εκ μέρους του θα ήθελα να πω ότι μετά από σχηνοτενείς διαπραγματεύσεις καταφέραμε να συμφωνήσουμε για ένα τελικό κείμενο για τη νέα αυτή συνένεση. Και οι δύο συνεισηγητές θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς Λίντα και όλους τους κοιόδης για τη συνεργασία τους και για την πολύτιμη συμμετοχή τους σε όλη τη διαδικασία. Να εκφράσω επίσης την ευγνωμοσύνη μας προς τη Γραμματεία και την Νομική Υπηρεσία και φυσικά προ, για, προς το προσωπικό μας και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μας για αυτό το σημαντικό θέμα. Ξέρουμε ότι η εκρίζωση της φτώχειας και η καταπολέμηση των ανισοτήτων και τη διακριτικής μεταχείρισης αποτελεί τον πυρήνα της αναπτυξιακής μας πολιτικής, στο πλαίσιο αυτή τη νέα Πιστεύω ότι η δέσμευση αυτή που συνδέεται στενά με την Ατζέντα του 2030 και τους στόχους βιασμής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών θα αποτελέσει την πιο σημαντική πολιτική δήλωση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής και των κρατών μελών της. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία, συνάδελφοι. Δεν ε, προλάβουμε. Έχουμε κάποιες τροπολογίες και κάποιες προφορικές τροπολογίες στην ε, λίστα ψηφοφορίας. Μπορούμε να δούμε τις προφορικές, αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την προφορική τροπολογία 2 και την 1 της Μαρία Χόιμποχ, που είναι ίδιες. Α, να δοκιμάσουμε πρώτα τα μηχανήματα. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Να δοκιμάσουμε. Βάλτε τις κάρτες για να δοκιμάσουμε να δούμε κατά πόσο το σύστημα λειτουργεί. Has everybody voted? Not everyone has voted. Can everyone just test? Λοιπόν, δοκιμάστε τα μηχανήματα για να μην πάει μετά κανεί και λέει ότι δεν δουλεύει το μηχανήμα του. Ποιο έχει πατήσει κουμπί, δεν έχει κουμπί, ποιος. Ψήφισαν όλοι. Το ΕΛΚ έχει μία παραπάνω, ένα CVP λοιπόν, ένα ΕΛΚ μπορεί να τη βγάλει. Ωραία, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, προφορική 2 και τροπολογία 1 της Μαρία Χόιμποχ. Ε, ποιος είναι υπέρ, κατά, α, ε, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 4 Παρακαλώ κύριε Έγγελ. Να σας ενημερώσω ότι είμαστε κατά της προφορικής τροπολογίας 4 όπως και των 6 ε, και 7. Έχουμε ένσταση για αυτές, θα μπορούσαμε να σηκωθούμε και όρθιοι για να εκφράσουμε την ένστασή μας. Δεν ξέρω αν το θέλετε να το κάνουμε σωματικά ή απλά να το πούμε. Αυτό ισχύει για την, όλη την ομάδα του ΕΛΚ, ναι, ότι είχε ένσταση προς αυτές. Δεν μπορούμε λοιπόν, αν υπάρχει ένσταση από δύο παραπάνω μέλη, να ψηφίσουμε. Οπότε η προφορική τροπολογία 4 καταπίπτει. Πάμε λοιπόν στην 2 και 3 έχουν αποσυρθεί. Πάμε στην 5 προφορική. 5 υπέρ, κατά, εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 έχει αποσυρθεί. Είπατε ότι έχετε ένσταση επίση για την προφορική τροπολογία 6 και 7. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να τη ψηφίσουμε. Ωραία, προφορική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6, καταπίπτει, εφόσον 8 έχει εγκριθεί. Όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε. Συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε την 6. Ποιος είναι υπέρ της 6, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα λοιπόν Για τα προφόρη ε, προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ας ψηφίσουμε τώρα επί του συνόλου του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας Εγκρίνεται με 15, 0 και 9 αποχές. Να ευχαριστήσουμε τους συνεισηγητές τον κύριο Νόιζερ που λείπει και τον κύριο Βέντα. Ευχαριστούμε για τις προσπαθίες τους. Ευχαριστώ συνάδελφοι. I'll give, I'll give the meeting a few moments to clear now. Many people are leaving, so we don't start with noise on the next item. So I'll give people a few moments to leave. Okay, colleagues, we can now move on to next. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Εάν επιθυμείτε να ε, συνδιαλεχθείτε, μπορείτε να εξέλθετε από την αίθουσα. Έρχομαι στο θέμα υπαριθμών 9, που πρόκειται για γνωμοδότηση για άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή, την ΑΦΕΤ, για διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Συντάκτης γνωμοδότησής μας είναι ο κύριος Κούλογλου και υπάρχουν και τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θα την ψηφίσουμε αύριο το πρωί, ώστε ό,τι θέλετε θα πρέπει να το πείτε τώρα. Στέλιο, έχετε το λόγο. Νομίζω... Uh, uh, Sorry, colleagues, people, yeah, people can. Yeah, thank you. Yeah, uh... Πρόεδρε, Είμαι βέβαιος ότι αυτά που θα πω θα βοηθήσουν τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν αύριο. Εν πάση περιπτώσει. Θα είμαι συντομότατος. Είναι ένα παγκόσμιο περίπλοκο φαινόμενο η διαφθορά. Αυτό θεωρούμε εμείς και τονίζουμε βεβαίως τη σημασία της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Οι δε τροπολογίες στις τροπολογίες μάλλον τονίζουμε τα αποτελέσματα της διαφθοράς ως παγκόσμιου φαινομένου, την ανάγκη του αγώνα κατά της διαφθοράς που πρέπει να θεωρηθεί προτεραιότητα απέναντι και μάλιστα στα εμπορικά συμφέροντα Και ένα σημαντικό ζήτημα είναι η συμπερίληψη ρητρών για ανθρώπινα δικαιώματα που να είναι δεσμευτικές, ώστε οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και κοινωνικά και να αγωνίζονται και αυτές για την καταπολέμηση διαφθοράς στις συμφωνίες που κάνουν. Τα έχουμε συζητήσει και με τη Γραμματεία και με τον κύριο Αουστρεβίσιους που είναι ο ε, εισηγητής της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής και η δική τους έκθεση θα ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Λίντα Μακάβαν, πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέντε. Α, με συγχωρείτε, όχι, με συγχωρείτε. Ο κύριος Κόσορ. Κόσα, συγγνώμη, εσείς είστε πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Στην ε, γνωμοδότηση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μιλούμε για τρίτες χώρες. Η παράγραφος 6 της αρχικής γνωμοδότησης είναι σημαντική για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και θέλουμε ξεχωριστή ψηφοφορία γι' αυτό. Δηλαδή η γνώμη μα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί σε τούτη εδώ τη γνωμοδότηση. Εγώ έχω υποβάλει τρει τροπολογίες και τέσσερις συμβαστικές. Το Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει τις περισσότερες τροπολογίες. Όμως υπάρχουν ορισμένε που το Λαϊκό Κόμμα δεν θα μπορέσει να τις εγκρίνει. Πρώτα, υπάρχει μόνο έξι. Πιστεύουμε ότι η ευθύνη των εταιριών δεν εντάσσεται στο πεδίο της εφαρμογής αυτής εδώ της ε, γνωμοδότησης. Για την 18 θέλουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Παράγραφο 18. Το ζητούμε αυτό διότι η εκπαίδευση, η παιδεία είναι σημαντικά πράγματα, αλλά εδώ μιλούμε για τρίτες χώρες. Και πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να δεχθούμε μόνο το πρώτο μέρος της τροπολογίας 18. Για την 21 δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, όμως υπάρχει ευτυχώς άλλη τροπολογία με παρόμοιο περιεχόμενο που είναι η υπαριθμόν 20 και αυτήν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν την υπαριθμόν 20. Και πάλι, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να παραμείνουμε σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με το πλαίσιο εφαρμογής της γνωμοδότησης και να εξαιρεθούν αυτά τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση, δηλαδή όπως η τροπολογία 24 και 28 που αναφέρεται σε μηχανισμούς καταγγελιών σε σχέση με εμπορικές συμφωνίες. Και βεβαίως συγχαρητήρια και ευχαριστίες των συντάκτη της γνωμοδοτήσεως. Ελπίζω ότι αύριο θα υπερψηφιστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω κάποιοι άλλου συναδελφοί να ζητούν το λόγο. Έχουμε τον κύριο Ολιβιέ Λούι από την Digitefco που βρίσκεται εδώ. Ε, συγγνώμη, είστε κάποιος άλλος. Όχι, εγώ είμαι. Ο κύριος Λουί. Νόμιζα ότι ήταν κάποιος άλλος, συγγνώμη. Λοιπόν, ε, να πω την άποψη της Κομισιόν για τη συζήτηση αυτή. Θα πω διάφορα πράγματα που είναι ήδη γνωστά, απλά θα σας παρουσιάσω μια περίληψη των όσων κάνει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν. Ε, υποστήριξη προς κυβερνήσεις ε, για τις υποχρεώσεις τους, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη κτλ. Η διαφθορά δημιουργεί διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στις δημοσίες υπηρεσίες υπέρ όσων μπορούν να επηρεάσουν τις αρχές για δικό τους συμφέρον. Ε, οι οικονομικά και πολιτικά μενεκτούντες λοιπόν ως αποτέλεσμα της διαφθοράς ε, εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα δημόσια αγαθά και υποφέρουν από αυτό. Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατηγικής τη ε, χώρες εταίρους για την καταπολέμηση της διαφθοράς η Κομισιόν ε, ακολουθεί μια πολυτομιακή προσέγγιση που αποσκοπεί στην δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτό περιλαμβάνει η μεταρρύθμιση της δημόσιας διαχείρισης, ε, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ε, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τελωνικές μεταρρυθμίσεις η απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποστηρίζει όχι μόνο τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων, αλλά και των οργανισμών επίβλεψης ε, και ελέγχου όπως τα μέσα, οι καταγγέλλοντες, ε, η κοινωνία των πολιτών, ε, καθώς και τα θεσμικά όργανα και τα κοινοβούλια. Αυτά είχαμε να πούμε για, για την ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν εδώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θέλει να πει κάτι. Ένα γρήγορο σχόλιο για να συμπληρώσω τα όσα είπε ο συνάδελφο. Έχουμε ήδη εκφράσει την υποστήριξή μα προς αυτή την έκθεση και στο παρελθόν και σε άλλε συζητήσει. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να επανερχόμαστε και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Ένα πράγμα μόνο στο νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 έχουμε μια ειδική προτεραιότητα, δραστηριότητα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ε, στην οποία δίνουμε μεγάλη σημασία στο πλαίσιο μια συνολικής ε, δράσης ε, ενίσχυσης των φορέων που συμμετέχουν και συνεργαζόμαστε μαζί τους και με την Κομισιόν για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Να υπενθυμίσω ότι τώρα μελετάμε την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης, ε, την ενδιάμεση αναθεώρηση, η οποία θα δημοσιευτεί τέλη Ιουνίου. Σίγουρα λοιπόν θα ξανασυζητήσουμε τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και σε αυτό το πλαίσιο. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Um, thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Κύριε Κούλογλου, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι. Όπως είπα συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Τώρα, α, για το επόμενο θέμα. Ναι, είναι εδώ το ε, αρμόδιο άτομο. Α, είστε εδώ. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τώρα θα περάσουμε ε, στο σημείο 10. Είναι αυτό που ονομάζουμε Global Gag Rule, ο κανόνας της παγκόσμιας φήμωσης, η Μέγγενης. Καλέσαμε άτομα από την Επιτροπή Γυναικών, από την Επιτροπή Προϋπολογισμού, Δικαιωμάτων να συμμετάσχουν σε αυτή την συζήτηση. Ο Ντόναλτ Τραμπ εξελέγει τον Ιανουάριο και αποφάσισε να, να, μην, να μην οι, οι ΜΚΟ οι οποίες έχουν χρηματοδότηση αμερικανική που δίνουν ε, συμβουλές ε, και υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες στις γυναίκες για τις αμβλώσεις ε, να, να απαγορεύεται να το πράττουν. Είναι κάτι που εμείς παρακολουθούμε στενά. Μήπως θα μπορούσε πρώτα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μας δώσει τη θέση της Νομίζω λοιπόν η κυρία Γκαρσία Περές έχουμε εδώ μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα θέλαμε ε, να πούμε ότι συμφωνούμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίδεται να μιλήσω για αυτήν τον παγκόσμιο κανόνα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι ε, μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια σε ολόκληρο το κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών και να προωθεί την ισότητα μεταξύ των φύλων και το δικαίωμα των γυναικών και κοριτσιών να αποφασίζουν ελεύθερα μόνες τους ποια προτεραιότητα δίνουν. Αυτή είναι προτεραιότητά μας στην υπηρεσία μας. Βεβαίως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τους στόχους χωρίς τη συμμετοχή των γυναικών μπορούν ε, οι ζωές ε, των νέων, των νέων γυναικών να σωθούν αν υπάρχει προστασία των ε, δικαιωμάτων των ατόμων να έχουν πλήρη έλεγχο για θέματα που σχετίζονται με την σεξουαλικότητά τους και στη σεξουαλική αναπαραγωγή και να μην έχουν να υποστούν καταναγκασμό και βία. Η δεσμεύση υπάρχει στα προγράμματα και στην πολιτική την αναπτυξιακή σε σχέση με την αναπαραγωγική υγεία, την εκπαίδευση, την σεξουαλικότητα, τις υπηρεσίες. Τώρα, σε σχέση με την ερώτησή σας, τις ανησυχίες μας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πανεισαγωγή του κανόνα αυτού της παγκόσμιας μέγενης και τελικά σε σχέση με τους στόχους, το στόχο μείωσης της ε, θνησιμότητας της μητρικής. Οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια στις στοχότερες χώρες του κόσμου υποφέρουν πολύ και υπάρχει κίνδυνος η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δεκαετίες για τις, τα δικαιώματα των γυναικών να χαθεί αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα πρέπει να παίξουμε έναν ρόλο για να βοηθήσουμε τις γυναίκες, τις οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι και μια προτεραιότητα, είναι ευθύνη μας και είναι μέσα στην εντολή που έχουμε. Η απειλή είναι πραγματική ε, και επίσης ε, σημαντική θα, σημαντικό θα είναι και το χάσμα το χρηματοδοτικό η κοινωνία των, κοινωνίες των πολιτών και άλλες ε, διεθνείς οργανώσεις αναλύουν ε, την, την, τον αντίκτυπο και, την, ε, και ποια θα είναι η καλύτερη προσέγγιση. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε με στεναρότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των γυναικών και νέων κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο και να προλάβουμε την βία, την σεξουαλική και κατά του γυναικείου φύλου, η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να προσπαθεί να κάνει περισσότερα διαφορετικά με, με, με καλύτερο στόχο, στοχοθετώντας κυρίως για τις πιο, τα πιο τροτά στρώματα της κοινωνίας, τις γυναίκες και διερευνώντας τρόπους να δράσουμε ε, διαφορετικά και γι' αυτό θα θέλαμε τις δικές σας ιδέες σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση κατατέθηκε από πολλούς. Θα ρωτήσω Ίσως την κυρία Ιντεβέλντα αν θέλει να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή της. Στο μεταξύ έχουμε λάβει και γραπτή απάντηση εντός της προθεσμίας και γι' αυτό τη βάλαμε και στην ημερησία διάταξη, το θέμα δηλαδή. Παρόλο που βεβαίως χαίρομαι για την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τις αρχές που προωθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά έχω το, το, ε, το αίσθημα ή την αίσθηση ότι δεν αρκούν αυτά τα πράγματα. Όταν λέτε ότι βασικά παρακολουθούμε την κατάσταση και μελετούμε τις επιπτώσεις, σκεφτείτε ότι ίσως είναι πια και πολύ αργά για πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές. Όπως είπατε, τα σχετικά εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο. Θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει πολύ ταχύτερα και ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση για την δημιουργία ενός ταμείου. Αυτό ήταν τότε δυνατό, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες ανταπόκρισης στη διάθεσή της και αυθόρμητα από ένα μέρος των χωρών μελών. Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ να περάσει, τόσο πολύ χρόνο να περάσει. Πρόκειται για επίγουσα κατάσταση όχι μόνο διότι επανέρχεται ο νόμος της Μέγενης, αλλά και επεκτείνεται. Θα είναι λοιπόν τεράστιες οι επιπτώσεις, όπως αρέσει τόσο huge, όπως αρέσει τόσο πολύ να λέει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ η ομιλήτρια που είναι στην ρίζα του κακού αυτού. Μιλήσατε για τις αρχές που οδηγούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να αναλάβει τις δράσεις αυτές, τα έλεγε και στην επιστολή του Σεπτεμβρίου 2015 που έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μας δεσμεύουν οι όροι του gag rule μεταξύ αυτών και η ρήτρα εμπιστευτικότητα. Σωστή αυτή η επιστολή, αλλά δεν είναι το ίδιο σαν να εφαρμόζεται ενεργά τις αρχές αυτές, διότι ο κόσμος επιτόπου πρέπει να γνωρίζει, να αντιληφθεί, να δει ότι όντως ισχύουν οι αρχές αυτές, ότι όντως υπάρχει χρηματοδότηση ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Και αν η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφαρμόζει ενεργά την πολιτική αυτή, ε, δεν ωφελεί και πολύ. Ελπίζω πραγματικά το ζήτημα να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη, ίσως να προβλεφθεί άλλη συζήτηση ή ψήφισμα ή κάτι σχετικό, αλλά θα θέλαμε πράγματι να δούμε μια πιο στέρεα απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι το οποίο να ξεπερνά την απλή παρακολούθηση ή αξιολόγηση των επιπτώσεων. Και αν δράσετε, θα έχετε την πλήρη υποστήριξη τουλάχιστον τη δική μου πολιτική ομάδα, αλλά νομίζω και τη πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ. Κάτι και μετά ο Σάρλ Γκέρεν. Πολύ λίγα έχω να προσθέσω στα όσα είπε η Σόφη. Μιλούμε βεβαίω για ορισμένες από τις πιο ευάλωτες γυναίκες και νεαρές κοπέλες σε ολόκληρο τον πλανήτη και πραγματικά αισθάνομαι βαθύτατη ε, θλίψη όταν ακούω, ερευνούμε και αναλύουμε τις επιπτώσεις ε, στην ουσία δηλαδή ένας κλασικός τρόπος κολυσιεργίας. Όπως είπε και η Σόφη, πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά. Πρέπει το χέρι βοήθειας που τίνει η Ευρώπη να φτάσει μέχρι τις κοπέλες και τις γυναίκες αυτές να γνωρίζουν ότι είμαστε στο πλευρό τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπόθηκαν τα ουσιαστικά από τις δυο συναδέλφους μου τα οποία υποστηρίζω πλήρω. Προσπαθούμε να βάλουμε τέλο σε μια παράλογη κατάσταση ή τουλάχιστον να αναπαλύνουμε λίγο αυτή την παράλογη κατάσταση. Αυτό ο παγκόσμιος κανόνας μέγενη, ε, όπως εκτελείται, όπως εφαρμόζεται, μα οδηγεί σε καταστάσεις ε, αποτρόπε ε, και παράλογες. Ας δούμε την περίπτωση μιας, ενός γιατρού που εργάζεται σε μια ΜΚΟ, σε μια περιοχή σειράξεων και υπάρχει μια γυναίκα τη οποία η ζωή μπορεί να σωθεί μόνο εφόσον τη παρασκευθούν οι απαραίτητε φροντίδε για μια άμβλωση και ο λόγο γιατρό βρίσκεται ενώπιον διλήμματο. Είτε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανόνα μέγενης, δηλαδή το απαγορεύεται να δράσει, διότι θα του κοπεί η χρηματοδότηση ή θα σκεφτεί τη χρηματοδότηση της ΜΚΟ του και σε αυτή την περίπτωση δεν θα κάνει τίποτα. Ή αν δράσει θα του κοπεί η χρηματοδότηση. Αυτό είναι παράδεκτο. Αυτό μας οδηγεί σε καταστάσεις ε, που έχουμε ξαναδεί. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για παρόμοιους λόγους η κυβέρνηση Μπούς είχε στερήσει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τους πληθυσμούς ε, ε, για, από χρηματοδοτήσεις σημαντικές ε, βάσει προσαρμογών του Ταμείου για τους πληθυσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είχαν βοηθήσει αμβλώσεις στην Κίνα. Το BBC εκείνη την εποχή είχε κάνει μια έρευνα για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν συνέβαιναν αμβλώσεις στην Κίνα ε, για την πολιτική αυτή του ενός παιδιού, όπως είχαν πιστέψει οι Αμερικανοί, και χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά αντισταθμίστηκε με κάποιον τρόπο το κενό αυτό χρηματοδότησης ε, από τα Ηνωμένα Έθνη. Και εδώ έχουμε μια παρόμοια περίπτωση. Είναι επίγον και πρέπει επίγοντος να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη. Η πρωτοβουλία αυτή του Τραμπ ελπίζω να έχει την ίδια επιτυχία με τα όσα έχει πει και κάνει στον τομέα της άμυνας και σε άλλους τομείς. Γιατί ε, βοηθά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τίποτα άλλο δεν βοηθά τόσο πολύ την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, γιατί σε τελική ανάλυση οι 28 χώρε, οι περισσότερε από αυτέ, αντιλαμβάνονται ότι πάμε ευθεία πάνω στον τοίχο. Οπότε από αυτή την άποψη πιστεύω ότι ο Τραμπ θα μπορέσει μια χαρά να λάβει το επόμενο βραβείο ο Καρλομάγνου. Ε, αυτό ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον για όσους θα πούνε οτιδήποτε στο Twitter. Ε, κυρία Μαριάν Πέτη, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζουν βάσει ποιων κριτηρίων θα παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια η οποία χρηματοδοτείται από του χρήματα των φορολογουμένων τους. Το ίδιο δικαίωμα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι πρέπει να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. Η άμβλωση δεν είναι μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού, ούτε πρέπει να προωθείται έτσι. Αυτό αναφέρεται σαφώς στο πρόγραμμα δράσης για τους πληθυσμούς ε, ε, των Ηνωμένων Εθνών και στη διακήρυξη του Πεκίνου. Θα πρέπει να ξέραμε ότι οι αμβλώσεις απαγορεύονται στο 8% των Αφρικανικών χωρών και τα κίνητρα για τη χρηματοδότησή της ε, αμβλώσης παραβιάζουν την νομοθεσία. Από την άλλη, πρέπει να αναλογιστούμε ποιος είναι ο στόχος μας. Η χρηματοδότηση των οργανισμών οικογενειακού πραγματισμού δεν αποτελεί υποστήριξη της δημόσιας υγείας η υγεία των γυναικών ε, δεν λαμβάνει καμία βοήθεια. Έτσι δεν διασφαλίζεται πόσιμο νερό ούτε τροφή, πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποιος ανθρωπιστικός οργανισμός λαμβάνει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πού πάνε αυτά τα χρήματα, γιατί εγώ δεν θέλω τα δικά μου χρήματα ή τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να χρηματοδοτούν παράνομες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ζοφκό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να συμμετάσχω στη συζήτηση και όπως είπε στην συνάδελφος Μαριάννα Πετή, θα ήθελα επίσης να ξέρω ε, πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια στις αφρικανικές χώρες αν καταλήγουν στο κράτος αντί να χρηματοδοτούν τις ε, αμβλώσεις, δεν πρέπει να εκπαιδεύονται οι γυναίκες ε, και να υπάρχει μια πρόληψη από τις μικρές ηλικίε. Νομίζω λοιπόν ότι οι περισσότερες συζητήσεις μας εδώ ε, στο Κοινοβούλιο, σε αυτήν την Επιτροπή για τις Αμβλώσεις, νομίζω ότι το κάνουν ε, ομιχλώδες όλο το θέμα. Τι γίνεται με την εκπαίδευση των γυναικών, με την ε, πρόληψη. Δεν είναι μόνο τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Είναι ντροπή που μερικά από αυτά τα θέματα ε, χρησιμοποιούνται έτσι για χειραγώγηση. Γιατί δεν επενδύονται περισσότερα χρήματα ε, για ψυχολογικές συμβουλές, ε, για πρόληψη συγκρούσεων, πρόληψη γενοκτονίας. Είναι λυπηρό να δει κανείς ε, ότι, ότι υπάρχει τέτοιο χάσμα ίσως σχετικά με την χρηματοδότηση της άμβλωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που λαμβάνετε υπόψη τις αξίες των χωρών αυτών, εκεί όπου δίδεται η βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν γνωρίζω όλους τους συναδέλφους. Είμαι νέο μέλος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μέλος ε, της Επιτροπής, της Επιτροπής ΦΑΜ, θα ήθελα να αντιδράσω στα όσα είπε η προλαλή σας, αν δεν γνωρίζετε ε, πώς ξοδεύονται τα χρήματα για ανθρωπιστικές βοήθειες ε, ή από πού προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, αν εξετάσετε τις δαπάνες, τις εκθέσεις των οργανώσεων IPPF, θα δείτε ότι επενδύουν τα χρήματα αυτά σε πάρα πολύ μεγάλη ε, ποικιλία τομέων, την ε, πρόληψη του AIDS, τα θύματα των ακροτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Έχουν γίνει πάρα πολλά, πάρα πολλά καλά ε, και βεβαίως αν ε, κοπούν αυτές, αυτή η βοήθεια από τις, Ηνωμένε, από τις θα γίνουν βιασμοί. Ε, βία θα υπάρξει, είναι σκάνδαλο. Με αυτήν την παγκόσμιο κανόνα της φήμωσης, της Μέγγενης, το είδαμε και προηγουμένως το 2004, και οι επιπτώσεις δεν ήταν μόνο αρνητικές ως προς την πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις, αλλά για την υγεία, την ε, μητρική, την πρόληψη του AIDS και ε, ε, μία από τις επιπτώσεις που δεν θέλουμε αλλά υπάρχει είναι ότι ο αριθμός των αμβλώσεων αυξήθηκε μετά την εισαγωγή του, του κανόνα αυτού. Θα πρέπει να δούμε τι είδους πολιτικής θα πρέπει να έχουμε για να υπάρχει μια κατάσταση όπου οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά της αναπαραγωγής και σε ασφαλείς ανβλώσεις με εκπαίδευση σεξουαλική. Υποστηρίζω το σημείο αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε το θέμα αυτό και υπάρχουν προτάσεις για μια, ανάλοψήφισμα ψήφισμα στην Ολομέλεια. Για δείτε τι γίνεται με, το πώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστούν χρήματα που χάθηκαν και τι κάνει και η Ευρωπαϊκή Επίτροπη και εμείς στην δική μας Επιτροπή θα λάβουμε απόφαση για να παρακολουθούμε το θέμα. Σοφίτ Βέλτ, ε, θες, ναι, ναι, πολύ σύντομα στους ε, δύο συναδέλφους που έλαβαν το λόγο προηγουμένως. Διαφωνούμε ε, σχετικά ε, διαφωνούν για το δικαίωμα σε ασφαλείς αμβλώσεις ε, και εγώ καμιά φορά, αλλά δεν είναι κάτι παράνομο, δεν είναι παράνομο. Αυτό είναι καθιερωμένο, υπάρχει σαφής πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι είναι μαύρο και τι είναι άσπρο. Είναι ανήθικο να μην βοηθούμε τις γυναίκες. Βεβαίως Πρέπει οι γυναίκες να εκπαιδεύονται, να ενημερώνονται. Αυτό, πρέπει να... Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις στερείται από το θεμελιώδες δικαίωμα να αποφασίζουν για τα δικό τους σώμα. Δεν αποφασίζουμε εμείς για τα σώματά τους. Δεν αποφασίζουμε για τα σώματα αυτών των γυναικών ή το δικό μου σώμα ή το σώμα κάποιας άλλης. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Εδώ μιλάμε για την πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξοδεύονται για αυτό το σκοπό. Η μόνη μου ερώτηση είναι τι αντίδραση θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το χάσμα αυτό, το κενό χρηματοδότησης λόγω της διεύρυνσης του παγκόσμιου κανόνα Μέγγενης. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό αυτό που λέει η Κομισιόν. Δεν λέω να κάνουμε κάτι παράνομο, να κάνουμε κάτι το οποίο είναι νόμιμο ε, και το οποίο θα πρέπει να επιταχυνθεί για να βοηθήσουμε τις γυναίκες που βρίσκονται σε απόγνωση σήμερα ως αποτέλεσμα αυτού του κανόνα. Όχι στο, μετά από πολλές εκθέσεις, αλλά σήμερα. Και τελικά δεν ξέρω πόσα κράτη-μέλη αποφάσισαν για αυτήν την She πρωτοβουλία. Ε, νομίζω θα έπρεπε να συγκεντρώσουμε όλους αυτούς τους πόρους και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει, να δράσει με αποφασιστικότητα και γρήγορα. Δεν νομίζω ότι θα λύσουμε τις διαφορές μας για τις αμβλώσεις. Η Επιτροπή μας Ανάπτυξης και η Επιτροπή Γυναικών θα έχουν μια κοινή έκθεση για εφαρμογής ε, σχετικά με το πρόγραμμα δράσης ε, ε, σχετικά με την ισότητα των φύλων για να υποστηρίξουμε τις γυναίκες μέσα στο πλαίσιο του αναπτυξιακό. Εδώ θα δούμε την όλη σειρά των δραστηριοτήτων. Ε, και πώς ξοδεύονται τα χρήματα για την εκπαίδευση των γυναικών των κοριτσιών. Δίνω και πάλι τον λόγο στην κυρία Βόφκο και στην κυρία Πετιέ. Ε, ναι, βεβαίω, κυρία Πρόεδρε. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Επειδή εγώ προέρχομαι από περιοχή που υπήρξε περιοχή σύραξη, ξέρω τι σημαίνει βιασμοί γυναικών σε περίοδο πολέμου τι μήνυμα θα στείλουμε σε αυτές τις γυναίκες που απέκτησαν παιδιά τότε ότι έκαναν λάθος. Δεν είναι ότι διαδίδουμε ότι λαμβάνουμε εμεί αποφάσεις ε, για τις γυναίκες αυτές χωρίς να τους δίνουμε το δικαίωμα. Εγώ λέω ότι αυτός εδώ ο θεσμός να συζητά πώς θα επενδύσει περισσότερα για να βοηθήσει οι γυναίκες να βοηθήσουν τους αυτούς τους. Αυτό έπρεπε να κάνουμε και όχι το να σκοτώνουν ζωές να τραυματίζει κανείς μια ζωή δεν βοηθάει κανέναν. Είναι εύκολο να σκοτώσει κανείς. Κατά την άποψή μου πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην παιδεία, στην ψυχολογική υποστήριξη, στην ε, κοινωνική φροντίδα, σε ε, αντιμετώπιση του μετατραυματικού στρες. Αυτά πρέπει να υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να επενδύει περισσότερα στις αμβλώσεις. Εγώ υποστηρίζω τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστούμε κυρία Πίτη. Να ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει χρηματοδοτικό κενό. Τα χρήματα αυτά καταβλήθηκαν σε οργανισμούς που ασχολούνται με οικογενειακό προγραμματισμό. Δεν εξαφανίστηκαν, υπόθηκε λάθο ε, κάτι τέτοιο. Τα κονδύλια αυτά υπάρχουν και θα τα λάβουν οργανισμοί που προωθούν ε, την υγεία γυναικών και παιδιών. Η πολιτική αυτή ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. Ε, παρόμοια ακούσαμε κάποια λάθος πληροφορίες εδώ. Ότι οι αυλώσεις ε, σώσουν τις ζωές των μητέρων και ότι αυτές περιλαμβάνονται σε αυτή την πολιτική. Αυτό δεν αληθεύει. και δεν περιλαμβάνεται φροντίδα μετά την άμβλωση. Οπότε θέλω οι συναδέλφοι να προσθέσουν σωστές πληροφορίες στη συζήτηση αυτήν. Αν λοιπόν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί δεν τηρούν την ομοθεσία των χωρών στις οποίες αναφερόμαστε και δεν πραγματοποιούν παράνομες αμβλώσεις, δεν θα υποστούν ζημία από τον κανόνα αυτό του Global Gag. πρόεδρος, η DigiDevco θα μιλήσει τώρα. Όχι, τη συζήτηση αυτή θα την κάνετε άλλη στιγμή, σα παρακαλώ. Έχουμε τον κύριο Πάλεφ από την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, ο κύριο Γιάννη Πάλεφ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να απαντήσω. Αλλά και εγώ θέλω να επαναλάβω ότι η Κομισιόν ε, συμμερίζεται ε, την ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις ε, του κανόνα αυτού της Μέγγενης για γυναίκες και για νέες γυναίκες ε, στο πλαίσιο διαφορών υπηρεσιών ε, και του κοινωνικού προγραμματισμού και το κατά πόσο θα ε, υπονομεύσει την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε θέματα υγείας, βελτίωση της υγείας και μείωση της ανεπιθυμητής μητρότητας. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία για τα δικαιώματα των γυναικών υπάρχει κίνδυνος να χαθεί. Όπω είπαν οι Επίτροποι Μιμίτσα και Στυλιανίδη, οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ δεν πρέπει να καθοδηγούνται από αυτά που κάνουν οι άλλοι ή που έχουν πάψει να κάνουν. Πρέπει να βασίζονται σε κοινέ ευρωπαϊκέ προτεραιότητε. Τώρα, όσον αφορά το pledging, την υπόσχεση, το να υπόσχεται κανεί χρήματα για κάτι είναι μία πτυχή μόνο. Η πιο δύσκολη δουλειά είναι ο προγραμματισμό και η υλοποίηση, ώστε τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν σωστά και όχι απλά να καλύπτουν κενά λόγω του περικοπών από τους Αμερικανούς. Θα πρέπει να αποτελούν κομμάτι μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και του σχεδίου δράσης της ατζέντα που έχει εγκρίνει η Κομισιόν. Όπως είπε ο Επίτροπος Μέμιτσα, δεν είναι αντί κάτι, αλλά προ ε, υπέρ των γυναικών η προσέγγιση αυτή. Σημειώνουμε ότι ναι υπάρχει καθυστέρηση, ότι δεν είναι αρκετά γρήγορο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η περικοπή δεν έχει συμβεί ακόμα. Τα σημερινά προγράμματα εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται και το σχέδιο εφαρμογής ε, ε, του αρμόδιου υπουργού στις Ηνωμένες δεν θα τεθεί αμέσως εφαρμογή. Ε, θα μπορούσαμε να δράσουμε και πιο γρήγορα βέβαια εμείς, αλλά ε, αυτό μπορεί να υπονομεύει τη δράση μας. Τώρα όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, ναι, ε, ε, έχουμε αιτήσεις εκθέσεις για τις δαπάνες των χρηματών των φορολογουμένων. Μπορεί κανείς να δει ε, τι έχει λάβει ο κάθε οργανισμός ε, από άψη Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Τώρα για την νομιμότητα φυσικά της αναπτυξιακής βοηθείας ε, εμείς πάντα δράμε βάσει συμφωνημένων ευρωπαϊκών πολιτικών όπως της Ευρωπαϊκής Συνένωσης για την Ανάπτυξη. Αυτό αποτελεί δεσμευσή μας ε, και στο πλαίσιο τη διεθνού διάσκεψη για του πληθυσμού και την ανάπτυξη των ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέτρο που σχετίζεται με τι αμβλώσει εντό του συστήματο υγεία μπορεί να καθοριστεί μόνο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και η χρηματοδότηση της Κομισιόν δεσμεύεται από τις αρχές αυτές και από τη νομοθεσία της ε, χώρας εταίρου. Ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Κάθη Περές, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, εν συντομία να ότι και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τι ίδιε ανησυχίε με αυτέ των συναδέλφων. Τόσο η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχουν υποστηρίξει την πρωτοβουλία και τι αρχικέ υποσχέσει, όπω είπε ο συναδελφό μου. Άλλο είναι το να κάνουμε υποσχέσει και να τι θέλουμε, και άλλο είναι το πώ προγραμματίζουμε τα χρήματα που ανέρχονται πλέον σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά υποσχόμενο ποσό. Είναι χρήσιμη συζήτηση όμω αυτή και καταλαβαίνω ότι θα συνεχίσετε από αυτά όσα ακούω τη συζήτηση αυτή. Άκουσα πολύ προσεκτικά τι απόψει τη Κομισιόν και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Θα συνεργαστούμε για την εφαρμογή. Φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι, οι ΙΠΑ δεν έχουν προβεί ακόμα σε περικοπέ όπω μαθαίνουμε. Δεν έχει περάσει ακόμα το Κογκρέσο αυτή, αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει στι ΗΠΑ, τι αποτελεί απλά ρητορική, τι θα εφαρμοστεί πραγματικά. Οπότε θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Να ευχαριστήσω του συναδέλφου που ήρθαν εδώ ε, και ειδικότερα οι προσκεκλημένοι από άλλε επιτροπέ. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για το σχέδιο δράση ε, και ελπίζω αυτό να οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη των γυναικών ε, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σα ευχαριστώ πολύ. αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Για σήμερα. Αύριο το πρωί στι 9 στην ίδια αίθουσα προβλέπονται ψηφοφορίε. Όσοι είστε αφιερωμένα μέλη τη Επιτροπή, έλθετε παρακαλώ με τις κάρτες σας.